Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και τους εσωτερικούς και τους επισκέπτες και τους μεμονωμένους βουλευτές έναν ένα. Είναι πάρα πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη, γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσω στην ώρα μου. Ε, ζητώ συγγνώμη, τι να κάνουμε αυτοί που καθυστερούν. Και θα ήθελα στην αρχή να έχουμε λίγο χρόνο να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα όσα συμβαίνουν ε, στην Ιαπωνία. Ιδιαίτερη θεομηνία, πρωτοφανή με πάρα πολλού νεκρού, ο δεν γνωρίζει πόσοι έχουν χάσει τη ζωή του και πόσοι ακόμα θα προσθεθούν στα θύματα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή και να θυμηθούμε τους ανθρώπους και να φέρουμε χρόνο στους ανθρώπους στην Ιαπωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις τώρα για την μέση διάταξη. Πρώτον, η έκθεση του συναδέλφου Ρέμιτ, που είναι το σημείο 15, αναβάλλεται για την Τετάρτη. Το έχουμε συζητήσει με τους ενδιαφερομένους, να το γνωρίζετε για να είστε εγκαίρους... Ε, παρόντες. Και ένα δεύτερο, αύριο το απόγευμα στις 5.30 θα έρθει ο κύριος Ότιγκερ, το συνεννοηθήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και το φιξάραμε σήμερα το πρωί. Θα έρθει ο κύριο Σότσιγκερ να μα μιλήσει για τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία και ε, τι συνέπειε θα έχει αυτό στην ευρωπαϊκή μα πολιτική. Αύριο στι 5.30 θα του κάνουμε και ερωτήσει, δηλαδή είναι μια επίκαιρη ώρα αυτή. Οπότε θα πρέπει λίγο να τελειώσουμε νωρίτερα στην ακρόαση. Λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη και από τον συνάδελφο Σούζα ε, Βάγνερ, αλλά ε, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε χρόνο στον κύριο Έτιγκερ. Θα, θέλαμε να τον έχουμε σήμερα, αύριο έχει συναντήσεις με εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία και από τις διοικήσεις και μετά, αμέσως μετά θα έρθει σε εμά. Νομίζω είναι η καλύτερη χρονική στιγμή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε γιατί από πρώτο χέρι θα μάθουμε και αυθεντικά τα όσα συνέβησαν. Μέχρι τις 5.30 θα πρέπει να έχει τελειώσει η ακρόαση, έτσι να τη στριμώξουμε την μέσα διαταξή της. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι και απρόβλεπτα θα ήθελα να πω επίσης ότι η κυρία Γιόρδαν Σίσελη είχε ένα τύχημα, γι' αυτό θα απουσιάσει αυτή την εβδομάδα, οπότε η ακρόαση θα γίνει μεν, αλλά θα πρέπει κάποιος άλλος συνάδελφος να προεδρεύσει. Ε, τώρα προσπαθούμε να το οργανώσουμε, ε, να το αναβάλουμε, δεν γίνεται να το ματαιώσουμε, απλώς να ξέρετε γιατί αλλάζει. Ε, να σας πω επίσης ότι αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη, όπως σας ε, ε, πρότεινα με τις αλλαγές που σας είπα, να την εγκρίνουμε και για το δεύτερο ανακοινώσει του Προέδρου. Θέλω να σας πω ότι στις 22 Μαρτίου το απόγευμα 3 με 6.30 στον τέταρτο όροφο θα κάνουμε ένα εργαστήρι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε, στις 22 το πρωί για το ETS, ε, άλλη επιτροπή, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Ε, τους υποσχέθηκα ότι θα τα πω και εγώ. Όπως και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, βεβαίως καλό την ίδια Επιτροπή αυτή να έρθει στην ώρα που θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Οίττιγκερ για να ενημερωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και από πρώτο χέρι και η συνάδελφοι Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αυτά τα εισαγωγικά σχόλια ανακοινώσει του Προέδρου. Το Σαββατοκύριακο πραγματικά ήταν πλούσιο σε γεγονότα, σε θέματα που σίγουρα θα μας ε, απασχολήσουν πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, τις εργασίες σήμερα και περνάμε στο σημείο 4, ε, ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Τσίσεστερ κάνει τη γνωμοδότηση, θα του δώσω πρώτα το λόγο και μια παρατήρηση μόνο θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να προσπαθήσετε να επικεντρωθείτε στις ομιλίες σας, να τηρείτε το χρόνο σας, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Να δείξετε κάποια πειθαρχία σας παρακαλώ πολύ. Είμαστε ε, κρίσιμη επιτροπή, σημαντική επιτροπή στο χρόνο που μας δίνουν θα πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ο Τσάρλς, έχεις το λόγο λοιπόν. Um, uh, θα ήθελα να στηρίξω ανεπιφύλακτα αυτά που είπατε προηγουμένως ε, σχετικά με το ότι πράγματι έπρεπε να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή για ε, αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία. Αυτά που με απασχολεί λιγάκι είναι... Εγώ είμαι αρμόδιος και για το σημείο 4 και για το 3 και για το 4 που έχουν σχέση με την προστασία των δεδομένων. Ε, το 3 είναι προστασία των δεδομένων και το 4 είναι το σημείο ενίζα. Θεωρώ λοιπόν ότι και εδώ πρόκειται για την προστασία των δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, ε, πράγματι έχουμε ε, πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα για αυτό το θέμα. Η αρμόδια επιτροπή επιθυμεί να προχωρήσουμε με την έκθεσή της και γι' αυτό ε, εμείς καταρτήσαμε ένα άτυπο έγγραφο εργασίας. Ζητώ συγγνώμη που είναι μόνο στα αγγλικά. Ε, θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τη γραμματεία για το ότι με υποστήριξε και πολύ γρήγορα υπέβαλε αυτό το έγγραφο. Ε, κυρίως για να το λάβουν υπόψη τους οι συνάδελφοι. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό τομέα της ε, δημόσιας πολιτικής. Ε, πρόκειται για ένα τομέα που βεβαίως και έχει να κάνει με την ελευθερία του ατόμου. Το θέμα της προστασίας των είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι έχω και ιδιαίτερο συμφέρον να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, γιατί όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, και εγώ ελέγχω τα δεδομένα με βάση την, το Μητρό του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία δεδομένων. Πρόκειται δηλαδή για μια νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να επηρεάζει και μένα προσωπικά. Κατά τα άλλα, ε, θα προσπαθήσω και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει ορισμένα θέματα. Και ε, θεωρώ ότι μετά την ανταλλαγή απόψε μπορούμε να προχωρήσουμε σε γνωμοδότηση, σε σχέδιο γνωμοδότησης. Το κοινοβόλιο λοιπόν συζητάει ένα θέμα το οποίο ετέθη Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει η έννοια της ε, ιδιωτικότητας, ε, υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και υπάρχει και η αρχή της ε, λογοδοσίας. Δεν είναι και τόσο πρωτότυπη η αρχή αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει τίθεται εδώ σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Εκείνο λοιπόν που θα να πούμε σε αυτό το έγγραφο εργασίας είναι ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες, κυρίως με την ευρύτατη έννοια. Δηλαδή, κυρίως όταν μιλάμε κάτι το οποίο πρέπει, το οποίο πρέπει να οριστεί με σαφήνεια στην νομοθεσία. Είπατε, Πρόεδρε, ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και εγώ δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες ε, σε αυτό το έγγραφο εργασίας. Ε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έχω κάποια αντίδραση από τους σκιώδεις ηγητές και μετά πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε γνωμοδότηση. Πάντως, θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πριν κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες ε, ε, θα επιβαρύνουν το φόρτο εργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, επιτιδευματιών γιατί αν επιβαρύνουμε περισσότερο τον έλεγχο των δεδομένων, αυτό πρέπει κανείς να το αιτιολογήσει. Πρέπει να υπάρχουν αποχρόντες λόγοι, γιατί ε, θα είναι ιδιαίτερη και επιπρόσθετη της ε, των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόζεκτο. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρε και με μεγάλη μου χαρά περιμένω τις αντιδράσεις των συναδέλφων και των σκιωδών εισηγητών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τσουκαλάς, παρακαλώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για το πολύ καλό έργο που έχει κάνει στο έγγραφό του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, επισημαίνει αρκετά σημεία στο έγγραφό του και γύρει διαφορετικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε όπως ε, η ασάφεια του ορισμού του ιδιωτικού βίου, κάτι που πρέπει να επιληθεί και μέσω της νομοθεσίας, το θέμα της λογοδοσίας, και επίσης το πώς αποθηκεύονται τα στοιχεία σε διαφορετικές βάσεις και σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Πρέπει λοιπόν να κοιτάζουμε ποιος είναι υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων και ε, ποιος, ποια δικαιοδοσία Εδώ μιλάμε για, ένα, για 1250 γιγαμπάιτ ε, προσωπικών δεδομένων συνολικά και ανακάτοικο του πλανήτη. Υπάρχει τεράστια αύξηση και ανάπτυξη και οι εταιρείε στο διαδίκτυο έχουν ε, την ευθύνη της, προστασίας των προσωπικών δεδομένων οπότε πρέπει να τις παρακολουθούμε. Η προστασία του ιδιωτικού βίου είναι ένας αγώνας δρόμου. Θα γίνει ψυχρός πόλεμος του 21ου αιώνα. Όμως τα θεσμικά μας όργανα δεν διαθέτουν πάντοτε την απαραίτητη ευελιξία για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Χρειάζεται λοιπόν εδώ ένα ευέλικτο πλαίσιο για να προσαρμοστεί η νομοθεσία για να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα και οι συστάσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στι καινοτόμε εταιρείε που θέλουν να παράσχουν υπηρεσίες σε εταιρείε, να δώσουν τέτοιε υπηρεσίες προστασία των προσωπικών δεδομένων η έννοια του ιδιωτικού βίου ε, ε, ήδη αναφέρεται. Εμείς ως νομοθέτες όμως δεν θα πρέπει να το δούμε από τη μηχανική μόνο πλευρά και των ε, υπευθύνων της πληροφορικής, αλλά και από κοινωνική πλευρά. Η προστασία από τους κινδύνους κατά του ιδιωτικού βίου για τους συμπολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι στοιχεία που τα χρειαζόμαστε. Οι προγραμματιστές λοιπόν των υπολογιστών θα πρέπει μαζί με τους νομοθέτες να λάβουν υπόψη τα στοιχεία του ιδιωτικού βίου για να υπάρχει μια ε, αρμόζουσα συμπεριφορά και εκτός διαδικτύου και εντός. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Τσάρλς για την έκθεσή του προσέχει πάντα υποδειγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί βλέπουμε από τη μια τις προσδοκίες και από την άλλη την εκπλήρωση αυτών. Δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Από τη μια έχουμε το Wikileaks ε, που το δοξάζουν και το υμνούν όλοι ότι να βγουν όλα να είναι δημόσια και ε, πέρα από κατηγορίες για κατασκοπία ή ε, παραβίαση του ιδιωτικού βίου. Από την άλλη αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική έχει καταστεί πλέον η ιδιωτική σφαίρα. Και αντικειμενικά θα πρέπει αφενός να προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα από τη μια και από την άλλη έχουμε το Wikileaks και καλείται ο νομοθέτης να ε, βολιδοσκοπήσει αυτή τη φαιά ζώνη για να καταλάβει πού είναι η πραγματική δύναμη Πολλά συστήματα έχουμε ήδη, όπως το ΕΜΑΣ, με θελοντική πιστοποίηση ε, για τους ε, επιχειρηματίες και κυρίως ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εθελοντικά θα πρέπει να παραμείνουν στην πιστοποίηση και να το υποστηρίξουμε. Αλλά τώρα δεσμευτικές και υποχρεωτικές ρυθμίσεις και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, επόπτες προσωπικών δεδομένων, κινδυνεύουν να προκαλέσουν μεγάλο κόστος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερο προσωπικό μοιραία, οπότε μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ε, Ευχαριστώ. Ως σκεώδης θα στηρίξω με την έκθεσή σας, αλλά θέλω να κάνω και κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ της ιδέας των επιγραμμικών και μη δεδομένων. Διότι δεν είναι το ίδιο δικηγόρο και γιατροί όπως οι εταιρείε ε, προϊόντων πληροφορική. Και οι εταιρείε αυτές δεν είναι το ίδιο με, με, τους, με ιστοτόπους. Δεν μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τους κανόνες σε όλους αδιακρίτως. Και αυτό και στο χρονικό περιθώριο που θα κατακρατούν, θα κατακρατούν τα δεδομένα πριν τα σβήσουν. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε όλοι κατά νου. Έπειτα υπάρχει ανάγκη, όπως είπατε και ο ίδιος, για μια σωστή, ένα σωστό ορισμό της έννοιας του ιδιωτικού βίου. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι τα ιστότοπα, οι ιστότοποι, όπως γενικότερα το διαδίκτυο, όλα τα προϊόντα του διαδικτύου πρέπει να εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό, τον σέβονται. Τον ορισμό του privacy by design. Είναι μια πολύ σαφής ιδέα που όμως θα πρέπει να την ε, διατυπώσουμε και με τον κατάλληλο, τρόπο. Τώρα για την συλλογή δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών, εδώ είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ώστε οι εταιρείε να ξέρουν πώς θα συσκευάσουν αυτά τα προϊόντα στην ουσία, πώς θα τα συναρμόσουν και θα τα στείλουν σε άλλες εταιρείε, σε ε, καταναλωτές. Πολλές φορές μάλιστα μετά από το πέρασμα κάποιου χρονικού διαστήματος, υπάρχουν και περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά επανέρχονται. Πολλές εταιρείε αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν τεράστιες βάσεις δεδομένων και από νομικής άποψη αυτό φαίνεται για την ώρα να είναι καλυμμένο. Θα πρέπει λοιπόν και την αγορά και την πώληση των προσωπικών δεδομένων να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο ποσοστό ηχνηλασιμότητα. να μπορεί να παρακολουθηθεί πορεία, να ξέρει κανείς δηλαδή σε ποιον απεστάλλει ένα προσωπικό δεδομένο, τι ώρα, ε, σε ποιο, ε, ποιος, ε, ο ελεκτή, μάλλον θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να υποβάλλεται και σε νομική λογοδοσία. Επίσης θα πρέπει να εργαζόμαστε σε, ομα... ομαδικό... σε ομαδική λογική ώστε να μπορούμε να δούμε ένα τρίτο μέρος πώς έχει λάβει κάποια δεδομένα. Εδώ λοιπόν για περιπτώσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μηνυμάτων από το Facebook, επειδή έχουμε λάβει τόσα πολλά, φαίνεται ότι είναι ζωτική σημασία και για τους ίδιου, και ότι πρέπει και εμείς να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτού του είδους το συντονισμό. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Λάμπερτ. Θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω στην διακατεύθυνση όπως η προαλήσασα. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε μια παγίδα και η παγίδα αυτή αφορά κυρίως τις νέες οικονομικές δραστηριότητες ε, και ε, κυρίως ε, την ανάπτυξη, μια λέξη που είναι ακούγεται πολύ ευχάριστη σε την Επιτροπή. Εσείς αναφερθήκατε στο Facebook ε, και στην πώληση δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά νέων επιχειρήσεων που αυτό το καθιστούν ακριβώς το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Δηλαδή πουλάνε πληροφορίες για τους ε, τελικούς χρήστες, στους τελικούς χρήστες, οποίους αποβλέπουν. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Ε, τα μέτρα βέβαια αυτά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το επιχειρηματικό προφίλ ορισμένων επιχειρήσεων. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο αυτό. Εμένα με απασχολεί περισσότερο ε, το θέμα της προστασίας των δομένων και όχι το επιχειρηματικό προφίλ ορισμένων επιχειρήσεων. Αλλά πρέπει αυτό που σας είπα να το έχουμε κατά νου. Διότι, Charles, νομίζω ότι ε, είπες και εσύ αυτό που είπε και η προλαλή δηλαδή θέλουμε να υπάρχει κάποια οικονομική δραστηριότητα, αλλά και εγώ πρέπει να προσθέσω όχι με κάθε τίμημα, νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που μου άρεσε, Τσάλ, ε, ε, στο άτυπο έγγραφο εργασία σου, είναι ότι αναζητάς την ευκρίνεια των ενιών. Δηλαδή, στο σημείο που μιλάς ε, για την ιδιωτικότητα, αυτό για μένα είναι αρκετά σαφές. Και αν θέλουμε να νομοθετήσουμε, ε, θέλω η νομοθεσία να είναι σαφής ε, και να μην καλύπτει τα πάντα. Άρα καλό αυτό που προτείνεις. Το πρόβλημα που με απασχολεί περισσότερο είναι το ότι έχουμε διαπιστώσει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ότι όταν κανείς αναζητά εργασία αυτομάτως γίνεται έρευνα στο παρελθόν του υποψήφιου εργαζόμενου. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα το παρελθόν τους σε κάποια στιγμή να διαγράφεται. Και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να ε, ανατρέχει και σε δεκαετίες, ολόκληρες δεκαετίες ε, στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον για τους ιστορικούς, αλλά όμως για εμπορική χρήση ή για χρήση που μπορεί να βλάψει το άτομο, αυτό ε, δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να βρούμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε το παρελθόν να διαγράφεται. Δεν ξέρουμε αν αυτή την άποψη μπορούμε να την εντάξουμε στην έκθεση, αλλά εγώ προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, από την Επιτροπή δεν έχουμε κανέναν ακόμα. Ίσως ο Τσάρλς θέλει να λάβει το λόγο και πάλι. Παρακαλώ κύριε Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους ε, για τις πολύ επικοδομητικές παρατηρήσεις του. Και επιτρέψτε μου να φερτώ σε ένα-δύο θέματα. Καταρχήν, ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο cloud computing και πρέπει να σας πω ότι ε, συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες του. Πρόκειται πραγματικά για μια ε, νέα έννοια. Όσοι υποστηρίζουν το cloud computing μου λένε ότι η ασφάλεια θα πρέπει να αυξηθεί και όχι να μειωθεί με αυτήν την ε, τεχνολογία. Και εγώ δεν είμαι πεπισμένος, θα δούμε. Το θέμα είναι Πώς μπορεί κανείς ε, να διατηρήσει την προστασία των δεδομένων ε, σε ένα τέτοιο μέσο. Αυτό δεν είναι μόνο φιλοσοφικό θέμα, είναι κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ τον κύριο Ρουμπίχ για την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του προς τα σχόλιά μου για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος είναι υπέρμαχος ένθερμος υποστηρικτής των μικρομεσαίων, όπως και εγώ. Κυρία Κολάσκα, είπατε ότι είναι σημαντικό online να υπάρχει διαχωρισμός του online από το offline. Εγώ όταν άρχισα ε, να παρακολουθώ το θέμα ε, του Μητρώου Προστασίας Δεδομένων στον Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσα ότι πρόκειται μόνο για δεδομένα ε, που υπάρχουν με ηλεκτρονική μορφή. Αν είναι σε χαρτία, αυτά δεν υπόκεινται σε αυτή την νομοθεσία. Άρα δηλαδή υπάρχει κάποια δυνατότητα παράκαμψης και πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό. Να λέμε ότι θα πρέπει ε, η προστασία να ισχύει και για τα δύο μέσα. Βεβαίως ε, η διατήρηση της θρητικότητας, ε, το να είναι κάτι απόρριτο σε χαρτί, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από, από σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Και γι' αυτό λοιπόν αν κανείς ε, θέλει να ε, διαβαθμίσει ένα έγγραφο, γράφει πάνω-πάνω, ε, διαβαθμισμένο και το μπορεί να το διαφυλάξει ως απόρριτο. Ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό λίγο παραπάνω όταν θα συντάξουμε το κείμενο της γνωμοδότησης. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για την πώληση δεδομένων, γιατί αυτό σημαίνει ε, ότι τα εμπορευματοποιούμε. Ενώ εμείς εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για την προστασία των δεδομένων. Ε, πάντως, ε, ο Φιλίπ Λαμπέρ αυτό που είπε σχετικά με το παρελθόν, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ως παρατήρηση και πάρα πολύ πολιτικοί θα έλεγα, ε, θα προτιμούσαν βέβαια σε μεγάλο βαθμό να διαγραφούν κάποια στοιχεία από το παρελθόν τους. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι ε, αυτό είναι λιγάκι οξύμορο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Πάντως... Ε, στο μέλλον μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προστασία και η ιδιωτικότητα, τόσο πιο πολύ επιτρέπουμε σε κάποιους ε, να ξεφύγουν, ε, να καταφύγουν σε πράγματα που αλλιώς δεν θα τα έκαναν. Αυτό βέβαια απασχολεί περισσότερο τον τύπο. Πάντως ε, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη συνάντηση των σκιωδών και να συντάξουμε τη γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν πρέπει σε αυτή τη φάση να συμφωνήσουμε στο χρονοδιάγραμμα κύριε Πρόεδρε, αλλά αν θεωρείτε ότι πρέπει παρακαλώ ενημερώστε με. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Μάλιστα. Ε, μέχρι τώρα είμαστε εντάξει χρονικά. Στις 11 Απριλίου, όχι, 11 Απριλίου είναι Λίμπε, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, πότε. 13 Απριλίου για μας. 13 Απριλίου, προθεσμία, για τις τροπολογίες. Δηλαδή, μέχρι τότε θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις προτάσεις σας, παρακαλώ. Και στις 9 του μηνός Μαΐου θα ψηφίσουμε. Ωραία. Και τώρα, αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, ε, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θαυμάσια, στην Ενίσα. Ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Κανονικά, θα πρέπει να έρθει ο κύριος Βουταρέλη εδώ στο Προεδρείο. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Äh, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εάν συμφωνείτε, να ε, περάσουμε στο σημείο 4 της ημέρας τη διάταξης. Καλώς ορίζω καταρχάς τον κύριο Μπουταρέλη και ε, του δίνω στη συνέχεια το λόγο για να μας ε, κάνει την εισαγωγή στι συζητήσει μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι χαρά και τιμή για μένα η ευκαιρία που έχω να συμμετέχω στην Επιτροπή σας, συνεισφέρω κι εγώ και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για την πρόσκλησή σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, μια σύνοψη να κάνω μόνο και να ενημερώσω την ε, γνωμοδότηση που υπέγραψα στα τέλη του περασμένου έτους, λαμβάνοντας υπόψη και μια άλλη ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα συζήτηση ε, αρχές Μαρτίου στο ε, ο όργανο του συμβολίου στην αρμόδια ομάδα εργασίας που ασχολείται με τα ίδια θέματα. Ως Ευρωπαίος Υπόπτης Προστασίας Δεδομένων, εμείς αντιμετωπίζουμε ε, πολλούς διάβλους συνεργασίας με την ΕΝΙΣΑ για το έγκλημα στο κυβερνοχώρο, για τα ε, θέματα ασφαλείας ε, και το θέμα του privacy by design που μόλις αναφέρατε, αλλά και τις καλύτερες ε, διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες. Αυτό εξηγεί γιατί είμαστε τόσο ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα και γιατί υποστηρίζουμε τις προτάσεις για να εξασφαλίσουμε την πλήρη συνέχεια της ΕΝΙΖΑ αλλά και να ε, εξυγχρονίσουμε και την εντολή της και να ενισχύσουμε το τομέα δραστηριοτήτων της, αλλά και να διευρύνουμε το πεδίο το οποίο καλύπτει. Όλα αυτά ε, γράφονται πλήρως στη δυνατότητα που δημιουργεί για την ενίσα πλέον η συνθήκη της Λισαβόνας να συνεργάζεται όχι μόνο με αρχές και όργανα επιβολής του νόμου αλλά και με αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι λογική και φυσική σύγκληση μεταξύ της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων πλέον και ε, η ασφάλεια των δικτύων είναι πάρα πολύ συστηματική και πάρα πολύ σημαντική για την προστασία και των προσωπικών δεδομένων. Τρία είναι τα σημεία που θα ήθελα να σας αναφέρω. Το πρώτο φορά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το νομικό μέσο που επιλέγεται είναι κανονισμός. Παρόλο που τα θέματα που αφορούν ε, και τις ε, αρχές επιβολής του νόμου αλλά και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων διατυπώνονται κατά την άποψή μας πάρα πολύ γενικόλογα σε όλη την πρόταση αυτή. Και αυτό επιτρέπει ευρεία ερμηνεία του συγκεκριμένου κανονισμού. Δηλαδή, το άρθρο 3.1 ε, κάπα λατινικό ορίζει ότι ο οργανισμός μπορεί να διεξαγάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που τις έχει αναθέσει νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι παραθυράκι όμω που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λειτουργία ή προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Και σα συνιστούμε για να αποφευθεί κάθε νομική ανασφάλεια και ασάφεια, ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σαφής και μονοσήμαντο για το τι δραστηριότητες και τι καθήκοντα μπορεί να εκτελεί στο μέλλον ε, ο οργανισμό ΕΝΙΣΑ. Το δεύτερο, τι συνδρομή μπορεί να ζητήσει η ΕΝΙΣΑ ή κάποιοι τρίτοι από τον οργανισμό αυτό. Ε, και πάλι ο κανονισμός έχει κάποια αναντιστοιχεία ε, σε σχέση με το ποιος μπορεί να ζητάει συνδρομή από την Ενίσα. Παράδειγμα. 7, 15, 16, μερικές αιτιολογικές σκέψεις 18 και 36 της πρότασης, αν τις συγκρίνετε και κοιτάξτε και άλλα άρθρα όπως είναι το 2, 1, 3 και 14, ε, θα διαπιστώσετε ότι αφενός γίνονται αναφορές σε ευρύτερη συνδρομή, ενώ ε, κάποια άλλα άρθρα περιορίζουν τον τρόπο συνεργασίας ε, ανάλογα με την οργάνωση ή το φορέα που ζητάει τη συνεργασία. Εμείς θεωρούμε ότι η ΕΝΙΖΑ θα, ε, πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστούμε όλα τα γραφεία, οι φορείς, οι οργανισμοί, τα θεσμικά όργανα καθώς και τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή αλλά και την υποστήριξη του οργανισμού αυτού. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΝΙΖΑ να ε, ασκεί τις ε, δραστηριότητες της όπου χρειάζεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης πρέπει να είναι και πιο επιλεκτικός οργανισμός για να είναι και πιο αποτελεσματικός. μια τρίτη ενότητα ε, σχολείων που θα ήθελα να σας κάνω είναι οι βέλτιστες ε, τεχνολογικές δυνατότητες. Οποιοςδήποτε οργανισμός της Ένωσης, φορέας κτλ. Καθώς και εμείς, ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, Προσωπικών Δεδομένων, έχει ξεχωριστή αποστολή. Και θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στις νέες τεχνολογίες και στην ασφάλεια. Γι' αυτό θέλουμε να ε, ε, στεθεί στην πρόταση μια σύντομη αλλά σαφής διάταξη που να λέει ότι θα χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατότητες, καλύτερες τεχνολογικά δυνατότητες ο οργανισμός αυτός και να αποτελεί υπόδειγμα ε, και παράδειγμα προς για άλλους οργανισμούς. Για να είναι σε καλύτερη θέση να ε, εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία. Γιατί τα μέτρα ασφαλείας ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει από τον εαυτό του αυτός ο οργανισμός. Γιατί τα λέμε αυτά. Διότι θα πρέπει να γίνονται πάγιες και μόνιμες ανταλλαγές με τη βιομηχανία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αρχείο, ένα repository και να, να ενημερώνεται, να ανανεώνεται αυτό σύμφωνα ε, με την πρόοδο της επιστήμης και αυτό να γίνεται σε μια βάση διαλόγου ε, πολύ εντατική. Εδώ συνδέεται αυτό και με τους νέους στόχους και με το νέο αντικείμενο που έχει πλέον ο ΕΝΙΣΑ. Η πρόταση δεν ξεκαθαρίζει αν και κατά πόσο ε, στα νέα καθήκοντα του οργανισμού εντάσσεται και ο χειρισμός προσωπικών δεδομένων. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να ισχύει και αυτό, να ε, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και εδώ χρειάζονται ειδικά μέτρα και να τα σκεφτούμε και να τα λάβουμε. Γι' αυτό συνιστούμε ότι αν ο οργανισμός θα πρέπει, και από ό,τι φαίνεται αυτό ισχύει, να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ε, ως αρμοδιότητά του θα πρέπει ο κανονισμός πρώτον να το ορίζει, να το ρυθμίζει και δεύτερον να ορίζει και έναν τρόπο ευέλικτο που να επιτρέπεται η επεξεργασία ε, κάποιων δεδομένων, να λέμε όμως ποια είναι αυτά και με ποια εχέγγυα και ποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Επίσης, συνεργασία και διάβλη συνεργασίας, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Συμπερίληψη ε, των διαφόρων ε, αρχών προστασίας δεδομένων, πάγια συνεργασία δηλαδή με τον οργανισμό αυτό, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να είναι συγκεκριμένη η διάβλη για τη συνεργασία των μηχανισμών. Γι' αυτό συνιστούμε οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων να έχουν ένα συνομιλητή στον ΕΝΙΣΑ βάσει πάντα του γνωστού άρθρου 29 της ομάδας εργασίας. και μάλιστα σε μια ρήτρα ε, μη ανάμειξης, ή τυπής του, του Ευρωπαίου επόπτη δηλαδή. Και μια τελευταία πρόταση έχει σχέση με τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μνημόνιο ε, που επεξηγεί τον τρόπο εποπτείας το περιγράφει ε, αυτά πολύ ξεκάθαρα. Εμείς συνιστούμε αυτή την προσέγγιση, αλλά επιπλέον θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτά θα πρέπει να ελέγχονται και εσωτερικά, να εγκρίνονται εσωτερικά και να υπάρχει και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Αυτή είναι η πρότασή μας, υποστηρίζουμε σαφέστατα τους ε, στόχους και τους σκοπούς, απλώς εμείς επιζητούμε περισσότερη σαφήνεια στον κανονισμό και όντως γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο και πρόσφατα βρήκαμε και υποστήριξη από πολλά κράτη-μέλη στην προσπάθεια αυτή. Δεν σας ε, ενθαρρύνουμε να είστε υπερβολικοί στις λεπτομέρειες και υπερρυθμιστικοί. Είναι μια καλή ευκαιρία να ε, βελτιώσουμε τον κανονισμό με περισσότερη σαφήνεια, χωρίς όμως να επιβαρύνουμε πάρα πολύ με λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ε, οι συνάδελφοι θέλουν ε, να μιλήσουν ε, πολύ, αλλά παρακαλώ, ο κύριο Σουκαλάς πρώτος, για δύο λεπτά έκαστος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλη για την παρουσία του εδώ, αλλά κυρίως για το εξαιρετικό κείμενο προτάσεων που ετοίμασε σχετικά με τη λειτουργία του ΕΝΙΖΑ. Η μεγάλη εμπειρία που πλέον συγκεντρώνει ο θεσμός του Data Protection Supervisor του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τα ασαφή σημεία και να υποβάλει κατά τη γνώμη μου ορθές προτάσεις για την αποσαφήνισή τους, τις οποίες τόσο εμείς όσο και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τις προτάσεις του κυρίου Μπουταρέλη για την εξέλιξη του ΕΝΙΖΑ σε de facto πρότυπο βελτίστων πρακτικών, τόσο για την διαδικτυακή ασφάλεια και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όσο και για τη σχέση που πρέπει να έχει με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βοήθεια που θα πρέπει να τους παρέχει. Η ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω προς τον κύριο Μπουταρέλη έχει να κάνει κυρίως με το πώς πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο ορατός, πιο παιδευτικός ο ρόλος και η αποστολή του ΕΝΙΖΑ τόσο ως προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και ως προς τους πολίτες. Δεδομένου ότι η ασφάλεια των δικτύων και η προστασία των δεδομένων αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος αλλά και του ότι η ενημέρωση, η προσωπική ευθύνη, η αυτοπροστασία, η προστασία και η εκπαίδευση έχουν για μένα τη μεγαλύτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ασφάλεια των πληροφοριακών μας υποδομών. Σας ευχαριστώ. Ganz herzlichen Dank und Charles Chichester ist der Nächste. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλη για τα σχόλιά του, τα οποία πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ, ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικά. Και θα ήθελα απλά να του κάνω μία ερώτηση που έχει σχέση με τη δεύτερη προτεραιότητα που ανέφερε και που έχει σχέση με την παροχή βοήθειας και με την ε, ασυνέπεια Ποιος δηλαδή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια από την ΕΝΙΖΑ. Συμφωνώ μαζί του ότι όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΝΙΖΑ στο φορέα αυτό. Θα ήθελα όμως να μας πει και τη γνώμη του για τη σχέση που υπάρχει, που ακριβώς εφάπτονται ο ΕΝΙΖΑ με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, κατά την άποψή του πώ πρέπει να εξελιχθεί η περαιτέρω σχέση. Πράγματι αναγνωρίζω ότι εδώ υφίσταται ένα κίνδυνος, ένας ε, κίνδυνος ε, να κατακλειστεί αυτός ο οργανισμός με αιτήματα ε, για βοήθεια, για προγράμματα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο τομέα που έχει σχέση με την πληροφορία και την ασφάλεια του διαδικτύου. Πάντως σε γενικές γραμμές ο ιδιωτικός τομέας έχει ιστορικό καινοτομιών και αυτό μπορεί να βολεύει πάρα πολύ το φορέα. Αναφερθήκατε και αλλού στις βέλτιστες υπάρχουσες ε, τεχνικές. Ε, φαντάζομαι ότι μπορεί να ζητήσετε παντού αυτές τις τεχνικές. Ίσως μπορείτε λιγάκι να επεκταθείτε περαιτέρω στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ΕΝΙΖΑ και τον ε, ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπουταρέλη κατά πόσο θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πιστεύουμε ότι η ευελιξία που αναφέρεται στον προτινόμενο οργανισμό αναφέρεται σε πολλά σημεία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Βεβαίως όλοι μας ε, θεωρούμε ότι ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ θα είναι καλύτερος ε, στο μέλλον, κυρίως ως ε, κέντρο τεχνογνωσίας. Θα είναι ένα καινούριο δίκτυο που θα αφορά και τους ιδιώτες και το κράτος. Το επεξηγηματικό μνημόνιο το επόμενο μάλλον, αναφέρει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, ο ΕΝΙΖΑ, θα διαδραματίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Και από την άλλη, η ενημέρωση για παραβίαση ασφαλείας, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ε, μέσα ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τομέας του εγκλήματος εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, εκεί ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ μπορεί να ε, διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε άμεση σχέση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούμε ότι το τμήμα εκείνο του κανονισμού το οποίο έχει σχέση με αιτήματα συνδρομής ε, το σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα ε, να υπάρχει κάποια δυνατότητα επιλογής ε, χωρίς ε, παράλληλα να υπάρχουν και περιορισμοί. Τώρα, όσον αφορά την ενημέρωση για παραβιάσεις και για το πώς είναι δυνατόν να εισάγονται έγκαιρα λύσεις στο δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Και η έρευνα είναι ένας τομέας όπου θα έλεγα ότι η είναι απαραίτητο να υπάρχουν θεσμικές επενδύσεις. Δεν είμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε τον οργανισμό ΕΝΙΖΑ, απλά πιστεύουμε ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα σε θέματα προστασίας δεδομένων και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό ΕΝΙΖΑ για την ενημέρωση σχετικά με παραβίαση θεμάτων ασφαλείας και θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει ε, πλήρης ε, σαφήνεια εμείς θα θέλαμε να ε, στηρίξουμε όλο αυτό το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μήπως επιθυμεί παρακαλώ να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίως που δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή να ε, σχολιάσει όλο αυτό το θέμα, να σχολιάσει τη γνωμοδότηση σχετικά με την ε, εποπτεία για την προστασία δεδομένων. Οι προτάσεις του ΕΝΙΖΑ ε, παρελήφθησαν μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή κατά κύριο λόγο εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους ε, τις προστασίας του επόπτη προστασίας δεδομένων και να δει πώς μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν ε, στον τελικό κανονισμό. Θα ήθελα απλά να αναφέρω δύο θέματα, να τοποθετηθώ σε δύο θέματα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικά. Πολύ συχνά ε, πολλές προτάσεις ε, του επόπτη προστασίας δεδομένων ε, αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτά όμως ήδη έχουν ενταχθεί στον οργανισμό. Δεν αποτελούν τμήμα του κανονισμού της ΕΝΙΖΑ, ούτε εντάσσονται στην παρούσα και στη μελλοντική εντολή. Όμως παρόλα αυτά, αυτά εφαρμόζονται μέσα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, το οποίο είχε εντολή να εφαρμόζει ε, τους κανονισμούς ε, του οργανισμού ΕΝΙΖΑ και αυτά προβλέπονται και από τον εκτελεστικό διευθυντή του ΕΝΙΖΑ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή δουλειά του οργανισμού και για θέματα προσωπικού. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα να παραμείνουν όπως σας τα παρουσίασα. Ο κανονισμός να αφορά θέματα στο ανώτατο επίπεδο και οι λεπτομέρειες της προστασίας των δεδομένων ε, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Ίσως λοιπόν εδώ είναι σημαντικό ε, να ε, διευκρινιστεί ότι το ε, Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει και αυτό έναν εποπτικό ρόλο. Αυτό είναι σημαντικό για την εφαρμογή των κανόνων περί προστασίας δεδομένων. Τώρα, όσον αφορά σε προτάσεις για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον κανονισμό του οργανισμού, κυρίως με τα καθήκοντα του κανονισμού, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία από πλευράς ε, οργανισμού, έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να εκτελεί καθήκοντα που δεν θα έχουν άμεση σχέση με τα ε, με τις τρέχους εξελίξεις, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί ε, σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Βεβαίως εναπόκειται στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουν τι μπορούν να αλλάξουν ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπουταρέλη, λέει ο Πρόεδρος, θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τελευταία σχόλια. Απλά θα ήθελα να πω ότι ο στόχος μας ε, να είμαστε ευέλικτοι και φιλόδοξοι, αυτός ο στόχος δεν αντιβαίνει, δεν βρίσκεται σε αντίφαση απαραίτητα με την αναγκαιότητα να υπάρχει σαφήνεια σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Όλοι μας επιθυμούμε ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ να μπορεί να ε, συνδράμει καλύτερα την Κομισιόν, να διευκολύνει τα κράτη-μέλη και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να υπάρχει μια περισσότερο ε, διεθνής προσέγγιση, μια ε, ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια, τις βέλτιστες ε, υπάρχουσες τεχνικές και την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι πρέπει πια να ξεφύγουμε από την κατακαιρματισμένη προσέγγιση που υπάρχει από πλευράς ορισμένων κρατών μελών. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση για να συνδυάσουμε αφενός όπως σας είπα αυτό το φιλόδοξο στόχο και αφετέρου την σαφήνεια. Ο κύριος Τσίτσεστερ θέλει και αυτός να κάνει μία παρατήρηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχολιά της ε, ε, Πολύ σωστά είπε αυτά που είπε ο κ. Μπουταρέλη για τον οργανισμό ε, και πολύ σωστά αυτά λέξα μετά την πρόταση για την έντολη γιατί με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ζωή όλων μας. Ε, θέλω λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλη. Νομίζω ότι όλοι ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση. Ε, θέλουμε να δώσουμε στον οργανισμό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί και επιθυμούμε όλοι ε, να υπάρχει σαφήνεια στα υποανάληψη καθήκοντα. Η ε, παρουσίασή σα. ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, τουλάχιστον για μένα που είμαι ο εισηγητής του θέματο. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρο, και εγώ ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να τα επαλαμβάνουμε. Αυτά ευχαριστώ τον κύριο Πουτρέλη και του συναντέλφου και για τι ερωτήσει και για τι πληροφορίε. Αυτή είναι μια διαδικασία που χρειαζόμαστε ακόμα ή έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο. 26 Μαου, μια μήνυα ακρόαση, το καλοκαίρι θα γίνει μελέτη. Αυτό το θέμα θα επανέλθει στη συνεδρίασή μα και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν σημαντικό το ότι σήμερα ασχοληθήκαμε σε βάθο με το θέμα. Και κλείνει αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Καλώς. Έχουμε μπει σε γοργούς ρυθμούς και χρονικά πάμε καλά σήμερα. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι δύο χωριστά τμήματα, αλλά έχουν μεγάλη συνάφεια ως προς το περιεχόμενο του 7 ο πρόγραμμα πλαίσιο και για τα δύο θέματα. Το πρώτο, έχουμε ένα προσκεκλημένο. Καλώς ορίσατε.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 τον κύριο Ρόλφ Άνεμπεργκ, πρόεδρο τη Ομάδα Εμπεριγνωγωμών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Είναι κύριοι και κυρίε που μπήκαν στον κόπο να κοιτάξουν αυτά, να τα ελέγξουν, να τα αξιολογήσουν, να μα πούν τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον, τι ήταν καλό, τι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο, τι ήταν λιγότερο καλό. Σα καλωσορίζω και σα δίνουμε την ευκαιρία να μιλήσετε σύντομα. Να μα πείτε ποια είναι η ενδιάμεση αξιολόγησή σα και στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία οι συνάδελφοι να ρωτήσουν. It's please. Ε, <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά ο κύριος Άνερμπερκ. Είναι μια ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλησίου. Και το απόγευμα σήμερα θέλουμε να δούμε πώς έχει διοργανωθεί, πώς έχει διαρθρωθεί η αξιολόγηση, ποια είναι τα βασικά μας πορίσματα και να πούμε και δύο λόγια για τις συστάσεις και το τι προβλέπουμε για το μέλλον. Κατά πρώτον, Λίγα λόγια για το ιστορικό της αξιολόγησης αυτής. Στην απόφαση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο αναφερόταν ότι μια ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο το 2010. Επίσης, ορίζεται στην ίδια απόφαση ότι θα πρέπει να καλύπτεται ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο, ότι θα πρέπει να διενεργηθούν αξιολογήσεις σε ειδικού τομείς, όπως το, Συμβούλιο, το Ερευνητικό Συμβούλιο της Ευρώπης και σε την, ε, το μέσο διευκόλυνσης για την ε, κατανομή του κινδύνου, λόγου χάρη. Ε, την αξιολόγηση αυτή τη διενήργησαν 10 ανεξάρτητοι ελεγκτές. Είχαμε 7 συναντήσεις από πέρσι τον Οκτώβριο και η έκθεση απεστάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου. Δεν θα μπω στα βιογραφικά και τις λεπτομέρειες της στα διαδρομία του καθενό από τα μέλη τη ομάδα αυτή, όμω όλοι έχουν παρελθόν στα οικονομικά, στι πολιτικέ επιστήμε, στην ε, πυρηνική φυσική, στην ιατρική. Και έχουμε και εκπροσώπους της βιομηχανίας ακόμη, από μεγάλες εταιρείε και από μια μικρομεσαία επιχείρηση. Εάν δείτε τώρα την εντολή που ανατέθηκε στην ομάδα αυτή, συμπεριλάμβανε 7 σημεία, 7 ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα αν έχουμε πετύχει τους γενικούς στόχους. Δεύτερον, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο της επιπτώσεις του προγράμματος και τις πολιτικές του. Ποιος είναι ο ρόλος του εβδόμου ου προγράμματος πλαισίου σε ένα διεθνές ε, πλαίσιο. Και μετά μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί πολλά νέα μέσα προβλέπονταν σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο, αν τα νέα αυτά μέτρα είναι αποτελεσματικά. Έπειτα, πώς μπορεί κανείς καλύτερα να αντιμετωπίσει τις ε, κοινέ προκλήσεις και το γεγονός ότι η συνεργασία, ο συντονισμό παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν ε, στο 7ο για την αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Αν ε, ήταν επίσης εύστοχα τα ερωτήματα ήταν το ερώτημα. Ήταν ευρύ το φάσμα όπως βλέπετε και αυτό ήταν καλό, γιατί όσο πιο ευρεία είναι η εντολή, τόσο περισσότερα μπορεί να καλύψει κανεί. Αν είναι στενότερη, πιο περιορισμένη, πολλά μπορεί να μείνουν απ' έξω. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι τα σημαντικότερα ε, σημεία τη εντολή αυτή καλύφθηκαν στην έκθεσή μα. Τώρα είμαστε στα μέσα της διάρκεια του 7ου προγράμματος πλαισίου. Μπορεί λοιπόν κανεί να πει Μάλλον δεν είναι εύκολο να πει κανεί από τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτή τη έρευνα στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμω ήδη κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα στοιχεία που συλλέξαμε τώρα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα από ό,τι συνέβη στην αντίστοιχη περίπτωση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, είχαμε την αυτοαξιολόγηση και τις, ε, τις εκθέσεις των ερευνητικών κέντρων και επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, μπορέσαμε να μιλήσουμε και με τους παλίλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποιες ήταν οι εμπειρίες τους από την διενέργεια του και την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Όλοι πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας διαβεβαίω είχαν πάρει την ε, υπόθεση αυτή πάρα πολύ σοβαρά και πολλές μελέτες είχαν γίνει από διαφορετικές χώρες αλλά από και ανεξάρτητους ε, ελεγκτές ε, και επίσης ε, δημιουργήσαμε και πολλές συνεντεύξεις με πάρα πολλούς ε, συμπολίτες μας, ερευνητέ, επευθύνους οργανώσεων που συμμετέχουν στην έρευνα και ούτω καθεξής. Επίσης είχαμε ευρύτατες διαβουλεύσεις κατά το καλοκαίρι με διάφορους ενδιαφερομένους και στο διαδίκτυο είχαμε τουλάχιστον 500 απαντήσεις. Ήρθαμε σε επαφή και με τα εθνικά σημεία επαφής ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς που ασχολούνται με την έρευνα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσωπούν μια εκατοντάδε εκατοντάδες ε, υπευθύνων. Τα πρώτα αποτελέσματα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα το βασικό μας μήνυμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Το εβδομο πρόγραμμα πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αναντήρητα δίνει μια σοβαρή συμβολή στην ευρωπαϊκή επιστήμη και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής έρευνα και του ευρωπαϊκού χώρου έρευνα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Πραγματικά λειτουργεί, αλλά παραμένουν και κάποιε δυσκολίε για ορισμένε από τι πτυχέ τη εκτέλεση του προγράμματο. Κατά πρώτον, είναι σημαντικό να βλέπουμε τι θετικέ πτυχέ. Τι είναι καλό στο πρόγραμμα αυτό. Ε, ας δούμε τώρα ποια είναι τα δυνατά σημεία του προγράμματος. Είναι πολύ μεγάλο ε, έχει πρόσβαση για πάρα πολλούς ερευνητέ και έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Εάν δείτε το τμήμα της συνεργασίας του 7ου προγράμματος πλαισίου, Είναι ο μόνο τρόπο που προσφέρεται για την ώρα για να έχουμε διασυνοριακή συνεργασία μεγάλη εμβέλεια. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα έχει σοβαρέ επιπτώσει στο πρόγραμμα αυτό. Κάποιε φορέ η επιστημονική ποιότητα του 7ου προγράμματο πλαισίου έχει τεθεί σε αμφισβήτηση. Όμως, εμείς πιστεύουμε οπωσδήποτε ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Η αριστεία ε, έχει επιδιωχθεί τα μάλα. Και πραγματικά νομίζουμε ότι η ποιότητα εδώ είναι εξαιρετική. Για την κινητικότητα. Είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της έρευνας και έχουμε καταλήξει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη από το Marie Κιουρί για την ε, κινητικότητα και την κυκλοφορία των ερευνητών και επιστημόνων. Και επίσης από φέτος βλέπουμε και τι πρώτε σοβαρέ επιπτώσει στις επιστημονικές και ερευνητικές υποδομές. Για την διευκόλυνση, όπω είπα, αξιολογήθηκε ξεχωριστά, θεωρήθηκε αποτελεσματική. Και εδώ είναι σημαντικό το εξή Υπάρχει μια σαφής, ε, υπάρχει σαφής, σαφές αποτέλεσμα ε, για το πώς οι εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και η βιομηχανία μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν. Τώρα για τους τομείς. Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση στους εξή τομείς. Πρώτα απ' όλα για το διοικητικό άχθος. Αυτό θα το δούμε και αργότερα αλλά σε κάθε περίπτωση για πολλούς ερευνητές, για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ επαχθής η διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμα, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Κατά δεύτερον, η έρευνα είναι κάτι το ρηψοκίνδυνο συνήθως. Συμπεριλαμβάνει ένα τεράστιο ποσοστό κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι δυνατό να υπάρχει και αυτή η πιθανότητα αποτυχίας κατά νου. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την ισορροπία μεταξύ κινδύνου και εμπιστοσύνη. Η πίστη, η εμπιστοσύνη είναι καθοριστική σημασία για την έρευνα. Παραδείγματα. Πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί και γι' αυτό έχουμε προβλέψει το TRE, το ανεκτό ε, κίνδυνο εισφάλμα. Επίσης για την συμμετοχή των γυναικών. Αργούμε, καθυστερούμε αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο ποσοστό του 40%. Ε, επίσης για την συμμετοχή βλέπουμε μια μικρή πτώση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και γίνει και στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Όμως οι στατιστικές μέθοδοι όπως τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ε, οι στατιστικές λοιπόν δεν είναι αρκετά σαφείς. Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι με τα στατιστικά δεδομένα ότι υπάρχει αυτή η τάση από την πλευρά της βιομηχανίας. Υπάρχει λοιπόν ο σχετικό στόχο, αλλά ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Κάποιε νέε μέρημνε και ανησυχίε μα έχουν απασχολήσει. Πρώτα απ' όλα, ανάγκη για αποτελεσματικότερο συντονισμό της έρευνας μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ακόμη και αν το πρόγραμμα πλαίσιο θεωρείται τεράστιο, υπάρχει παρόλα αυτά εξίσου μεγάλος όγκος και ποσοστό χρημάτων, κονδυλίων και στα κράτη-μέλη. Ε, εδώ χρειάζονται τεχνολογικές πρωτοβουλίες, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά υπάρχουν και παράπονα. Μας λένε ότι οι διαδικασίες που προβλέπει το πρόγραμμα είναι περίπλοκες. Ή υπάρχουν προβλήματα για τους νεοεισαχθέντες, νεοεισαχθέντες το πρόγραμμα. Ένα άλλο νέο στοιχείο είναι το άρθρο 185 που δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμη αρκετά γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Και για τον κοινό προγραμματισμό το ίδιο. Επίσης, κάτι που μας ανησυχεί πολύ, σε πολλούς τομείς έχουμε χαμηλά ποσοστά επιτυχίας για το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο και επιτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 και για τα νέα κράτη-μέλη που δεν είναι πια τόσο νέα, είναι χαμηλότερα τα ποσοστά επιτυχίας για τους καινούριου παρά για τους παλιούς. Αλλά και κάποιοι από τους παλιούς έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Αυτό το συζητήσουμε τόσο ή για μακρόν. Ένα άλλο θέμα είναι ο χρόνος που υπάρχει για τη χρηματοδότηση Δηλαδή, το πότε υποβάλλει κανεί μια πρόταση, μια υποψηφιότητα και μέχρι πότε φτάνει να πάρει τη χρηματοδότηση στα χέρια του. Αυτό καταναλώνει ένα μεγάλο μέρο του 7ου προγράμματο πλαισίου και χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή από την άποψη τη διαχείριση. Τώρα, που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να οδεύουμε για το υπόλοιπο διάστημα εκτέλεσης του 7ου προγράμματος πλαισίου και του 8ου όμως πρέπει να επικεντρωθούμε στις μεγάλες όπως ονομάζουμε προκλήσεις. Κλιματικές αλλαγές, ανταγωνιστικότητα, γύρω στο πληθυσμό και ε, προμήθεια ενέργειας. Επίσης χρειάζεται μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τρίγωνο της γνώσης όπως έχει ονομαστεί. Δηλαδή και η εκπαίδευση να στην ερευνητική μας πολιτική. Εάν θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη ε, συμπερίληψη των ερευνητικών πολιτικών και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα φιλοσοφία και θα πρέπει με μια νέα ματιά να δούμε τη διεθνή διάσταση του προγράμματο πλαισίου. Θα πρέπει επίσης να πυκνώσουμε τις διασυνδέσει μεταξύ των βασικών υπευθύνων έρευνας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και αλλού. Έχουμε δέκα κύριες συστάσεις, αν διαβάσετε την έκθεση θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλες πολλέ, όμω εδώ έχω σταθεί στις πλέον σημαντικέ. Είναι σημαντικό Εάν θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους για την ένωση της ε, καινοτομίας και του χώρου έρευνας, να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό της έρευνας. Πρέπει να επικεντρωθούμε, να στοχεύσουμε σε λιγότερα ζητήματα, τις μεγάλες προκλήσεις που έλεγα προηγουμένως. Ιδίως εκεί που απαιτείται μια κρίσιμη μάζα. Δεύτερη σύσταση. Χρειαζόμαστε υποδομές υψηλής ερευνητικής ποιότητας. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και οι λεγόμενοι S3 ε, οδικοί χάρτες έχουν ετοιμαστεί. Όμως ε, θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθούν δραματικά οι υποδομές στα τελευταία στάδια του προγράμματο. Ω προ τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ε, στοιχεία ότι τα κονδύλια δαπανώνται ορθότατα. Βέβαια υπάρχει μια τάση δαπάνε να είναι περισσότερες προ το τέλο παρά στην αρχή του προγράμματο. Αλλά εδώ θα πρέπει να διατηρήσουμε σταθερό το επίπεδο χρηματοδότηση. Και αν περισσέψει κάτι τα τελευταία στάδια, να το διαφυλάξουμε για το επόμενο πρόγραμμα. Επίση, χρειάζεται μια καλά διαρθρωμένη στρατηγική καινοτομία και απλούστευση. Ε, όποιον και αν ρωτήσετε, όποιον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, εάν σα ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ω τώρα, θα σα πει τρία πράγματα. Απλούστευση, απλούστευση και απλούστευση θα ζητήσει. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο ζήτημα. Δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί τα προβλήματα να λύνονται με την απλούστευση την τεχνική την τεχνικό εννοούμενη. Χρειάζεται και στην, ε, στο επίπεδο τη λήψη αποφάσεων, το πολιτικό, η απλούστευση. Γι' αυτό λοιπόν για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα που ήδη διαθέτουμε ενώ για το 8ο, το επόμενο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση των ε, δημοσιονομικών κανονισμών. Κάτι που ούτως άλλως προβλέπεται. Επίσης πιστεύουμε σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ της ανάντη και κατάντι προσέγγισης, bottom-up και top-down, εκεί θα πρέπει να εξεύρουμε με πιο σωστή ισορροπία. Είναι δύσκολη ε, η προσπάθειά μας, διότι το περιθώριο συνεργασίας που έχουμε ως τώρα είναι περιορισμένο. Αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίε και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και στου ερευνητέ. Εάν το περιθώριο ήταν μεγαλύτερο, θα ήμασταν αποτελεσματικότεροι, πιστεύουμε. Υπάρχουν πολλά νέα εργαλεία, όπως σας είπα, που προβλέφθηκαν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και θα γνωρίζετε ότι είναι απλούστερο να δημιουργεί κανείς καινούργια πράγματα παρά να χρησιμοποιεί, να αξιοποιεί τα παλιά. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να χρειαστεί ένα μορατόριο, μια περίοδο πάυσης χρήση των νέων ε, εργαλείων μέχρι να αναπτυχθούν επαρκώς και να είναι και αρκετά καλά αποτιμημένα έπειτα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την συμμετοχή των γυναικών, διότι όπω είπα ο στόχο ήταν 40%, όμω είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Αν δείτε το συνολικό πληθυσμό των Ευρωπαίων ε, ερευνητών, φτάνουμε το 30% δύσκολα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταβάλει προσπάθειες για τα πάνελ, για τις ομάδες ερευνητών, όμως πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη αυτό και τα κράτη-μέλη. Επίσης, λίγα λόγια για τα κάτι μελη που δεν εκπροσωπούνται αρκετά. Δεν θα το λύσει αυτό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, όμως θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε καλύτερη συνεργασία και με τα υπεύθυνα ταμεία για να το επιλύσουμε αυτό. Έπειτα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι ανοιχτό στην διεθνή συνεργασία βέβαια, αλλά είναι πολύ λίγε οι προσπάθειε και πολύ διασκορπισμένε. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια σαφή στρατηγική, προκειμένου η διεθνή συνεργασία να συμπεριληφθεί σε όλα τα τμήματα του προγράμματο. Τέλο, Κάποια σύντομα σχόλια για το 7ο, για το 8ο, συγγνώμη, πρόγραμμα πλαίσιο. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό τώρα το αντικείμενο τη συζήτησή μα, όμω σύντομα θα γίνει αντικείμενο συζήτηση. Έχουμε λοιπόν κάποιε ιδέε και γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, ποια θα πρέπει να είναι η προσέγγιση. Θα πρέπει να έχουμε έμφαση στην βιομηχανία και περισσότερη διασύνδεση έρευνα με την κοινοτομία μεγαλύτερη συγκέντρωση στις μεγάλες όπω τις ονόμασα πριν προκλήσει, στρατηγικό επαναπροσανατολισμό τη διεθνούς συνεργασίας, πραγματικές αποτελεσματικές διασυνδέσεις μεταξύ έρευνα και καινοτομίας, αλλά και ενίσχυση τη έρευνα και τη κατάρτιση στην έρευνα. Επίση, βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Ε, η μερίσια διάταξη της έρευνας ε, θα μπορούσε να διοργανωθεί επίσης. Μιλάμε εδώ για θέματα αριστείας, ε, ανταγωνιστικότητα, η βιομηχανία εκεί γράφει την ημερήσια διάταξη και καθορίζει τις εξελίξεις και διάφορα θέματα που επιβάλλει η κοινωνία και διαφέρεται να ερευνηθούν. αυτά σταματώ εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, αυτέ ήταν οι πρώτε πληροφορίε εισαγωγή. Τώρα έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε πρώτα από τον κύριο Ντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια κύριε Άνερμπερκ είναι συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε και σα παρακαλώ να διαβάσει στου υπολείπου εμπειρογνώμονε τα συγχαρητήρια τη Επιτροπής μα, διότι το έγγραφο είναι πολύ σημαντικό αυτό και μα επιτρέπει να προετοιμάσουμε το ψήφισμα, την έκθεση πρωτοβουλία ε, με τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μα τη δική αξιολόγηση, τη θέση του Συμβουλίου και την ανακοίνωση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σα κάνω μερικέ ερωτήσει. Στην αξιολόγησή σα έχουμε την εκτύπωση ότι ε, ότι είστε πάρα πολύ στοχευμένοι στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, που είναι καλό για την εντολή σας αυτή, αλλά δεν επεκτείνεστε στη γενικότερη δημόσια έρευνα στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη. Όμως, μεγάλο μέρος της έρευνας διεξάγεται στα κράτη-μέλη. Και έχουμε λίγο την εντύπωση ότι, δεν θα έλεγα βέβαια, να φτάσω μέχρι να πω ότι δεν υπάρχει πιλότο στο αεροπλάνο, αλλά αυτός ο συντονισμός κράτος-μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται πάντα, θα άξιζε να γίνει και δεν έχουμε και αξιολόγηση εκ των υστέρων από αυτόν. Βλέπουμε την εντολή σα και την επιστολή σα που αναθέτει, δεν σα το έχουν ζητήσει. Είναι λογικό να μην απαντάτε. Αλλά έχετε καμιά αίσθηση να μα διαβιβάσετε ε, πώ συνεργάζονται τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την απλούστευση ευχαριστώ πάρα πολύ που μα υποστηρίζετε, διότι είναι πάγιο μέλημά μα και έτοιμά μα από την απαλλαγή του 2007 Επιτροπή η δική μας και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και χαιρετίζω την κυρία Καρβάλιο που έχει κάνει καταπληκτική έκθεση πάρα πολύ υψηλής ποιότητας γι' αυτό. Εσείς μιλήσατε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε και για το 6ο όμως ακριβώς υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα για την υπερβολική γραφειοκρατία και το διοικητικό φόρτο και ε, επιμένω για το μέλλον και τονίζω ότι θα πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι και απευθύνομαι στον άλλο πρόεδρο τώρα, τον κύριο Ρόιλ, γιατί δεν καλύψατε το θέμα ε, του κινδύνου και πώς επιμερίζεται αυτός θα κάνουμε άλλη συζήτηση εδώ για τον αντίστοιχο μηχανισμό, άλλη αξιολόγηση, δεν ξέρω, ρωτάω τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, η κυρία Ερτσόκ. Or somebody else who named Thanks, Chairman. I was... Herzog. <laughs> no, I was not sure that I applied in, in so early stages uh, certainly. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έπαιρνα το λόγο τόσο γρήγορα. Ε, πιστεύω ότι προηγούνται άλλοι. Μπα περιπτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας κύριε Αγμπερκ, και θέλω να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Ε, μερικές εξ αυτών ε, μοιάζουν με αυτές που αφορούν και τον κύριο Οντί. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος ε, πλαίσιο. Ε, βεβαίως πρέπει να μπείτε και πιο βαθιά. Ας πούμε, ε, χαμηλός δείκτης επιτυχίας σε, σε ορισμένους τομείς. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Είναι νέοι στο εβδόμο ο πρόγραμμα πλαίσιο ή είναι οι παραδοσιακοί τομείς. Το ίδιο ισχύει και για τον χαμηλό δείκτη επιτυχίας στις 12 χώρες σε σύγκριση με τις 15. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά από την πρώτη διαφάνεια που μας δείξατε, εγώ κατάλαβα ότι κανείς από τους 12 δεν ήταν παρόν στην ομάδα εργασίας. Ισχύει αυτό ή ήταν ε, επίσης παρόντες και ε, συνάδελφοι από τις 12 χώρες. Και κατόπιν, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και τα νέα έντυπα. Παρήματο χάρη, ε, αξιολογήσατε τα νέα έντυπα που να αφορούν στις ε, κοινοπραξίες και μας ενδιαφέρει αν είναι επιτυχημένες κοινοπραξίες ή όχι. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μορφή συνεργασίας ή μήπως είναι αποτυχημένη και πρέπει να ζητήσουμε κάποιες νέες μορφές και τέλος, σε αυτό που είπε ο κύριος Οντί, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δραστηριότητες του κράτους μέλους και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, να υπάρχουν καλύτερες ε, μετρήσεις. Ε, δεν έχετε να παίξετε μόνο κάποιο ρόλο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και στις δραστηριότητες των κρατών μελών για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην έρευνη και την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ που θα απαντήσετε σε ερωτήσεις μου και ευχαριστώ και που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Οντί, ε, μία σύντομη απάντηση αν θέλετε και η γραμματεία μου επισήμανε ότι το θέμα της, ε, του επιμερισμού κινδύνων αυτό συζητήθηκε εδώ πριν από κάποιες εβδομάδες. Απλά εγώ κάπως δεν άκουσα καλά. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούει κανείς εξωτερικές απόψεις από εξωτερικούς ε, συνεργάτες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν ορόσημο και επειδή είμαι και μέλος Επιτροπής Προπολογισμών, η αύξηση κονδυλίων του 7ου σε σχέση με το 6ο ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εσείς την αύξηση ε, κονδυλίων για το 8ο πρόγραμμα πώς την αξιολογείτε. Θα ε, υπάρξει αύξηση σε ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι θα μπορούσαν εκεί να χρησιμοποιηθούν ήδη οι πόροι, παραδείγματος χάρη τα αποτελέσματα από τις ε, δημοπρασίε για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, γιατί κατ' ουσίαν αυτές οι, αυτές οι ε, και οι διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν στόχο να διαπιστωθούν ε, αυτές, το επίπεδο των εκπομπών. Και κάτι άλλο, πώς βλέπετε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Τεχνολογίας από κοινού με το πρόγραμμα SIP ή επειδή πιστεύουμε ότι το, η καινοτομία πάει προς το 8ο πρόγραμμα, ε, θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα SIP Competition Implementation Program ε, το οποίο θα έχει ως στόχο ε, την καινοτομία να τη μεταφράζει, να τη μεταφέρει στην πραγματική οικονομία και στην παιδεία με στόχο η γνώση να επηρεάσει επί της ουσίας τα εκπαιδευτικά συστήματα και την παιδεία γενικότερα. Κυρία Ριέρα Μαδουρέλα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να αρχίσω με ευχαριστίες προς τον κύριο Άνερμπερκ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για την παρουσίασή σας και για την εργασία σας και εσάς προσωπικά και το συνάδελφο σας στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι εύκολο βέβαια να κάνει κανείς ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά για μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και ε, πριν ολοκληρωθεί το 7ο και πριν έχουμε την οριστική αξιολόγηση. Αναφερθήκατε σχεδόν στα πάντα εσείς, αλλά θα παρακαλούσα αν μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο σε κάποιους στόχους ε, που θέσαμε όταν ε, αποφασίσαμε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο και δεν ε, μπήκατε σε λεπτομέρειες. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έγινε στο πρόγραμμα για να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Από ό,τι φαίνεται η βιομηχανία συμμετέχει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν σε προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο, ιδιαίτερα στην καινοτομία ή σε ένα ειδικό πρόγραμμα για τη συνεργασία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιωτική συμμετοχή και ε, πώς έχουν εκμεταλλευτεί και πώς έχουν αξιοποιήσει τα μέσα και τα μέτρα, το GTI που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, και είπατε ότι υπήρξαν κάποια παράπονα, κάποιες καταγγελίες ή θέματα στόχων του 15% συμμετοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που και πάλι αναφερθήκατε παρόδο χωρίς να ε, μας ε, δώσετε την αξιολόγησή σας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να αφαιρθώ στους ανθρώπινους πόρους Αναφερθήκατε στις υποτροφίες Marie Curie, είναι πάρα πολύ σημαντικές όντως για την κινητικότητα των ερευνητών, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα αν ε, έχουμε καλύψει τους στόχους ε, ε, αύξηση του αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν. Η Ευρώπη είναι ελκυστικός προορισμός για ερευνητές τρίτων χωρών. Βοηθάμε τους νέους να ακολουθούν αυτή την επιστημονική σταδιοδρομία συμφωνώ και με τον κύριο Οντή που σας ρώτησε πώς αξιολογείται τη λειτουργία, αν βελτιώθηκε ή όχι, του συντονισμού μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και των κρατών μελών και μέχρι τις περιφέρειες και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη χρηματοδότηση. Συνεργάζονται. Ακούμε μερικά σχόλια για τα κοινοτικά κονδύλια ε, ότι αυτά δεν πιάνουν τόπο στην καινοτομία και στην έρευνα, αλλά το χρησιμοποιούν για να υποκαταστήσουν πολλές φορές ε, την εθνική χρηματοδότηση. Επίσης, πώς αξιολογείτε το συντονισμό, το αναφέρατε, αλλά δεν επεκταθήκατε με άλλα προγράμματα και άλλες κοινοτικέ δράσεις. Και επίσης, δεν ξέρω αν πετύχαμε τη ε, διεπιστημονική πτυχή αυτή τη συνεργασία των διαφόρων, τι γίνεται με τους κοινού διαγωνισμούς, της κοινέ προκήρυξεις. Ευχαριστώ. Ο ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση που την ε, βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Επειδή το θέμα της έρευνας είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας. Γι' αυτό πρέπει να επενδύουμε πάντοτε περισσότερο στην έρευνα και την κοινοτομία. Ιδίω για τους νέους, τους νέους ερευνητές. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό. πρώτο ερώτημα λοιπόν. Πώς να ευνοήσουμε την ε, εκπαίδευση των νέων ερευνητών, την συμμετοχή τους μέσω του προγράμματος πλαισίου. Δεύτερο ερώτημα που εμένα μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, με απασχολεί ιδιαίτερος. Η σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Το λέω γιατί είχα και μια άμεση προσωπική εμπειρία. Πολλές φορές είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, για να προσεγγίσουν ε, τα προγράμματα αυτά και να αποκτήσουν μια σχέση. Πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε ιδίω το τμήμα που αφορά την απλούστευση, όπως αναφέρατε. Κάποιες φορές οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, ακριβώ επειδή είναι μικρές, δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα προγράμματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξαναδούμε το σύστημα χρηματοδότησης. Διαδικασίες λογιστικές, πολλές φορές βλέπουμε αυτές οι διαδικασίες να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Και επίσης κάτι που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε περαιτέρω, να εμβαθύνουμε σε αυτό για να στηρίξουμε ακριβώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα ευνοήσουμε το κόστος σχεδιασμού ε, που αναλαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να μην τι επιβαρύνουμε περαιτέρω στα προγράμματα έρευνας όλα αυτά. Αυτά ως προς την απλούστευση και για να τελειώσω και να κλείσω η εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου ως σήμερα φαίνεται να είναι διασκορπισμένη μεταξύ πολλών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο κατακαιρματισμός περιπλέγεται στις καταστάσεις Εκεί που ακριβώς χρειάζεται όμως ομοιογενής και ενιαία εφαρμογή των κανόνων και διαδικασίες για να δοθούν τελικώς επιδοτήσεις ε, υπέρ της έρευνας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι δεν είναι απλώς επιθυμητό αλλά και απαραίτητο να βελτιωθούν αυτές οι διαδικασίες, να απλουστευτούν ώστε να μπορέσει να υπάρξει άμεση εκτέλεση και ευκολότερη πρόσβαση του εβδόμου προγράμματο προγράμματος πλαισίου ε, για λόγους που γενικότερα θα ευνοήσουν την καλή εκτέλεση του προγράμματος. Ευχαριστούμε κύριο Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Άνερμπεργκ για την εδώ παρουσία του. Σύντομες θα είναι οι ερωτήσεις μου. Ε, θα περίμενα, επειδή μου λείπουν τα στοιχεία πριν να αρχίσουμε να εξετάζουμε πολιτικές ή αξιολογήσεις του εβδομου ου προγράμματος, να είχαμε μια γενική εικόνα σε σχέση με την διεθνή θέση της ευρωπαϊκής έρευνας και τεχνολογίας και τις τάσεις που δεν φαίνεται να είναι ε, πολύ αισιόδοξε για την Ευρώπη, όπως ακριβώς αν κατάλαβα καλά και στο ε, σχέδιο που θα διαβάσουμε του κυρίου Οντή σε λίγο μας υπενθυμίζει. Αυτό το λέω διότι ε, έχουμε ενεξελίξει το όραμα του 2020 που διαδέχεται την αλίστου μνήμη στρατηγική της Λισαβόνας και ποτέ κανείς δεν μας εξηγήσει ποια είναι η πραγματική παγκόσμια θέση της ευρωπαϊκής έρευνας τόσο ως προς την χρηματοδότηση όσο και ως προς τα αποτελέσματα. Επομένως, θα ήμουν ευγνώμων αν ε, ίσως ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής έκανε ένα hearing κάποια στιγμή σε σχέση με τη θέση της Ευρώπης, σε σχέση με την παγκόσμια, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε έρευνα και τεχνολογία και τις προοπτικές του 2020 ή του 2025 όπως ε, δείχνουν και οι πρόσφατες μελέτες. Επίσης, στη δεύτερη και τελειώνω ερώτηση, ο κύριος Άνερμπεργκ είπε κάπου ότι τα κονδύλια εξοδεύονται ορθότατα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, η κυρία Καρβάλιο μας το έδειξε προσπαθώντας να βρει τρόπους για πλούστευση των διαδικασιών, όμως σε πρόσφατη ερώτηση που έκανα στην Κομισιόν μου απάντησε ότι δειγματοληπτική έλεγχη του 0,4% των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν απέδειξαν λάθη στο ύψος του 4%. Ελπίζοντας ότι το μοντέλο δεν είναι γραμμικό και ότι όταν ελέγξουν το 4% δεν θα βγουν λάθη 40%, σας υπενθυμίζω ότι στα 50 δις το 4% των λαθών είναι 2 δισεκατομμύρια. Άρα σας ερωτώ γιατί αποφαίνεστε ότι τα κονδύλια ξοδεύονται ορθότατα δεν έχω την ίδια αίσθηση. Ο Καβάλιο. Κύριε Καβάλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για αυτή την πολύ καλή παρουσίαση για το θέμα της απλούστευσης και την διάρθρωση του 7ου προγράμματος πλαισίου θα ήθελα να σχολιάσω. Για την απλούστευση, όπως είπατε, Έχουμε δύο σειρέ μέτρων. Πρώτον, αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρί να αλλάξει ο δημοσιονομικό κανονισμό. Και από αυτήν την ομάδα μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εφαρμόσει κάποια και πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε τρία συγκεκριμένα μέτρα απλούστευσης που θα προβλεφθούν. Υπάρχουν όμως και άλλα που μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάξει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου ή το σφάλμα και ο δημοσιονομικός κανονισμός. Ε, ούτε μάλλον ο δημοσιονομικό κανονισμό. Άρα για την έκθεση του κυρίου Οντί, και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, ε, για την έκθεση του κυρίου Οντί θα πρέπει να υποφεληθούμε τη ευκαιρία για να προτείνουμε μέτρα πλούστευση που δεν απαιτούν περαιτέρω αλλαγέ και σε άλλου κανονισμού. να εφαρμοστούν όσα διαθέτουμε ήδη στα χέρια μα, δηλαδή. Ήθελα να ξέρω και τη δική σα άποψη. Θα ήθελα να το αποσαφενίσετε, παρόλο που φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, για τη διάρθρωση του 7 προγράμματος πλαισίου. Νομίζω θα έπρεπε, καθότι έχουμε χρόνο ακόμη και κονδύλια, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, από όσα δεν πάνε καλά. Βεβαίω, από ό,τι φάνηκε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, είναι πολλά τα στοιχεία που πηγαίνουν καλά, οπότε να μην τα πειράξουμε, μην κάνουμε αλλαγέ ε, ω αυτόν τον σκοπό. Όμω, ό,τι είναι βελτιώσιμο, να βελτιωθεί. Και έπειτα ήθελα την άποψή σα για τρία πολύ σύντομα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ των μεγάλων, όπως είπατε, προκλήσεις και της ε, έρευνας της bottom-up. Ε, Βεβαίω υπάρχει το Ερευνητικό Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και τα προγράμματα συνεργασίας. Ποια είναι η άποψή σας για το να έχουμε κάποιο πρόγραμμα συνδυασμού των τεχνολογιών στο μέλλον. Κάτι που χρησιμοποιείται ήδη πάρα πολύ στον τομέα της ε, πληροφορίας, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, ICT. Υπάρχει εδώ περιθώριο για νέες ιδέες σε ό,τι αφορά τη διάσταση της συνεργασίας στο πρόγραμμα. Και δεύτερη ερώτηση. Άκουσα κατά τις διαβουλεύσεις περί απλούστευσης πολλά παράπονα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τη μια για την απλούστευση τα αναφέρατε στην εκθεσή σας τα περί απλούστευσης, αλλά και για το σχεδιασμό ε, του προγράμματος, ε, των καθεαυτών προγραμμάτων. Αυτά λένε βελτι... ευνοούν πολύ περισσότερο τις μέσες δομές, τα μέσα ερευνητικά κέντρα, τις μέσες ερευνητικές ομάδες που ως ε, διάμεση κάνουν κάποια πράγματα για λογαριασμό των ε, επιχειρήσεων. Ζητούν λοιπόν ένα σχεδιασμό τη πρόβλεψη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και τώρα για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, το τρίτο μου σχόλιο. Για να έχουμε και το βλέμμα στραμμένο προ την αγορά. Ήδη με τα πολλά ερευνητικά προγράμματα πλαίσια που είχαμε ω τώρα, βλέπουμε αξία να παράγεται όταν τα επιτυχημένα, οι επιτυχημένες ερευνητικές προσπάθειες μπορούν να εφαρμοστούν και σε επακόλουθα στάδια προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα καλά αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο να αξιοποιεί κανείς την καινοτομία. Πρέπει να υπάρχουν πλαίσια τέτοια προγράμματα που να επιτρέπουν ε, τα αποτελέσματα της έρευνας, οι θετικές επιπτώσεις να έρχονται και πιο κοντά στην αγορά. Για αυτήν την αξιοποίηση λοιπόν των άριστων αποτελεσμάτων της έρευνας, ποια θα ήταν η άποψή σας, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τα εκμεταλλευτούμε πλήρως. Η ε, κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Παρακολούθησα πάρα πολύ ε, στενά την αξιολόγηση, τη διάβασα επανειλημμένα και σας συγχαίρω για αυτή. Έχω κάποιες ερωτήσεις κανονικά να κάνω στον καθηγητή. Θα μπορούσατε να συμπληρώσετε λίγο την ενημέρωση για τα όσα τονίσατε ήδη. Παράδειγμα, μιλήσατε για τα μέσα και τα εργαλεία για την καινοτομία και για το μορατόριο, να μην δημιουργήσουμε άλλα πριν ευδοκιμήσουν αυτά που έχουμε. Δεν μας λέτε όμως για τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να κάνετε ένα βήμα παραπέρα και να δείξετε ειλικρίνεια και να το ρυψοκινδυνεύσετε κι εσείς, όπως λέτε ότι είναι ρυψοκίνδυνο το θέμα της έρευνας. Τι συμβαίνει. Εγώ είμαι υπέρ του να δημιουργήσουμε, να συνεχίσουμε συγγνώμη με τα μέσα που έχουμε, να μην δημιουργούμε νέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει προπαγάνδα και το λέει και flagship, εμβληματικές πρωτοβουλίες. Και τι θα πει αυτό και τι εστί καινοτομία για την Κομισιόν. Δεύτερον, Κάτι που μου λείπει από την αξιολόγησή σας είναι και πάλι για την καινοτομία και σχέση καινοτομία με την έρευνα. Μέγα τμήμα της καινοτομία έρχεται από το κράτος υποχρεωτικά, γιατί στην Ευρώπη πάνω από 70% των επιχειρήσεων είναι δημόσιες χωρίς να φαίνονται πολλές φορές. Γνωρίζουμε όμως ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι δημόσιες. Και στην Ισπανία ε, λέγεται Comtech, μια μεγάλη έρευνα που έγινε και το κράτος δεν αγοράζει καινοτομία, αγοράζει χρηματοδότηση. Για να μην το πάμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, ε, στις περιφέρειες ας πούμε ή σε ε, τοπικά νοσοκομεία δεν μπορούν να αγοράσουν τη τεχνολογία και δεν την εφαρμόζουν γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Άλλη ερώτηση. Και πώς συμμετέχει ο ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν συμμετέχουν ορισμένες χώρε ή είναι χαμηλή η συμμετοχή τους. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ε, στη χρηματοδότηση γιατί ο συντονισμός γίνεται στα οικονομικά. Όχι, θα πρέπει ο συντονισμός να γίνεται στην αριστεία, να είναι τα κριτήρια συμμετοχής κριτήρια αριστείας και να επιβραβεύονται ε, οι χώρες που τα εισάγουν αυτά. Ενώ συζητάμε τώρα για τα κονδύλια, για την περιφερειοποίηση, για την κατανομή. Ε, διαπραγματευόμαστε στο Συμβούλιο πόσα χρήματα θα πάρει κάθε κυβέρνηση ε, στη χώρα της. Ε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα θέματα της έρευνας. Το κριτήριο θα πρέπει να είναι ακριβώς η αριστεία. Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία συνδέεται με την προηγούμενη. Μιλούμε για τους ανθρώπινους πόρους. Με τα πανεπιστήμια τι γίνεται στην Ευρώπη. Και τελειώνω. Υπάρχουν χώρες όπου δεν λειτουργούν καλά τα μέσα υποστήριξης του 7ου Προγράμματος. Στη χώρα μου, την Ισπανία, οι διαγωνισμοί, οι προκηρύξεις αποκλείουν τον ιδιωτικό τομέα. Ε, τότε μετά πώς ζητάμε λεφτά από τους ιδιώτες, αν δεν τους επιτρέπουμε να ενταχθούν από την προκήρυξη του διαγωνισμού στα ερευνητικά προγράμματα. Μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν. Μεγάλα ιδρύματα αποκλείονται επίση ιδιωτικά. Αυτό τι σημαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια που αποκλείονται και θα μπορούσαν. Στις άλλες χώρες τι γίνεται. Αυτά, τελείωσε ένα πακέτο ολόκληρο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμσον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ε, ευχαριστώ και για την πολύ καλή παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πράγματι ε, θέσατε τον δάκτυλο στον τύπο των ήλων και μου άρεσε πάρα πολύ ε, το ότι καταλήξατε στο ότι η ευρωπαϊκή υπεραξία είναι πράγματι πολύ σημαντική γιατί πρέπει αυτή την υπεραξία να την προβάλλουμε στα ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, ε, συνδυάζεται όλα αυτά με τις ερευνητικές δομές, με τις δυνατότητες και τέλος και με την εθνική έρευνα, την έρευνα στα κράτη-μέλη. Ε, όμως, εκεί που κάτι αναζητώ είναι στο θέμα της ε, βελτίωσης. Εσείς μιλήσατε για το διοικητικό άχθος, αλλά όχι για περιορισμούς όταν μιλάμε για έρευνα. Στο Κοινοβούλιο, όταν μιλάμε για βιομηχανία, δεν μιλάμε κατ' ουσία για τη βιομηχανία, αλλά μιλάμε για την μεταποίηση. Και ελπίζω όταν ε, μιλάτε για οικονομία και βιομηχανία, εννοείται αυτό και όχι το, τη μεταποίηση. Το 75% απασχολείται σε αυτόν τον τομέα. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να βρει κανείς τη σχέση της βιομηχανίας με την έρευνα και μετά. Το θέμα το ε, διατομεακό, διακλαδικό. Εγώ έχω και εμπειρία, έρχονται ερευνητέ και διαμαρτύρονται, μου λένε ότι θέλουν να ασχοληθούν με τη νανοτεχνολογία στην Ευρώπη και παίρνουν τηλέφωνο το Business School της Κοπεχάγης για να τους πούν πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις. Το να καταρτήσει κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω αυτά που είπατε σχετικά με τις ε, μεγάλες προκλήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτά έχουν με τον γυράσκοντα πληθυσμό, ε, την ενέργεια, την παραγωγή εναλλακτικών ε, ενέργεια από εναλλακτικέ πηγές. Χρειαζόμαστε λοιπόν για να τα ερευνήσουμε όλα αυτά και τους κοινωνιολόγους. Πρέπει κανείς ε, να διατηρήσει την πολυεπίπεδη έρευνα και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αναπτύξουμε νέες δομές. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα προγράμματα. Εγώ δεν νομίζω ότι πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει χρειάζονται έρευνα, χρειάζονται τη μεταφορά γνώση ω αποτέλεσμα τη έρευνα. Και αυτό, αυτή, αυτός ο διάβλος ε, θα πρέπει να ε, δρομολογηθεί, να καταρτιστεί ίσως ως ένα κομμάτι της ε, τεχνολογίας ε, καινοτομιών. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχουν στήσει αρκετή το λόγο και ο κύριος Άρεμπερκ ε, θα ήθελε να δώσει και κάποιες απαντήσεις. Ίσως λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο... να εξετάζουμε ε, ταυτόχρονα και το επόμενο σημείο της μερικής διάταξης, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε το χρόνο για τις απαντήσεις. Ε, λοιπόν, ε, εξετάζουμε άρα και το επόμενο σημείο της μέση διάταξη. Ο κύριο Άρμπεκ, θα δώσει τώρα κάποιες απαντήσεις και μετά θα συνεχίσουμε και με άλλες ερωτήσεις. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρώτα απ' όλα προς τον εισηγητή, τον κύριο Ντί. Το πρώτο σημείο εδώ για τη σχέση των κρατών μελών και το τι κάνουν σε αυτό το τομέα μετά όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίω είναι άκρα σημαντικό όλο αυτό. Όπως ορθώς είπατε, εδώ στην εντολή μας δεν συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση όλης της ευρωπαϊκής έρευνας. Αυτό όμως που έχουμε δει ως τώρα είναι εάν η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή έρευνα και η ευρωπαϊκή καινοτομία μπορούν να ασχοληθούν με τις μεγάλες, όπως είπαμε, προκλήσεις, τότε είναι πιο εύκολο να βρεθούν διάβλη συνεργασίες των κρατών με, την, με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε τα κονδύλια, υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί, διαφορετικοί ορισμοί επίσης, όμως μεταξύ εβδόμου προγράμματος πλαισίου που συμβάλλει περίπου στο 5 με 15% της των συνολικών ερευνητικών δαπανών στην Ευρώπη, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη-μέλη καλύπτουν κάτι μεταξύ του 85 και 95%. Άρα προφανώς χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Χρειάζονται μέτρα και μέθοδοι και διαδικασίες προκειμένου όλα αυτά να λειτουργούν αποτελεσματικά. Κάποια τα διαθέτουμε ήδη από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε μικρότερης εμβέλειας προγράμματα. Έχουμε το πρόγραμμα έρευνα ΣΥΝ και το άρθρο 185 και την ιδέα του κοινού προγραμματισμού, του joint programming, δηλαδή για συγκέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε κάτι να φροντίσουμε να γίνει για τις μεγάλες προκλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό και για την αξιολόγησή μας και για το μέλλον. Να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Καταλαβαίνω επίσης ότι αυτό σας απασχόλησε και κατά τη σύνταξη της εκθεσής σας. Έπειτα μιλήσαμε για την απλούστευση. Νομίζω συμφωνούμε την ίδια άποψη έχουμε από τη Ουσίας Τονίζω όμως ξανά ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να το λύσουν οι υπάλληλοι και οι τεχνικοί. Εάν θέλετε να εκτελεστεί σωστά και ο δημοσιονομικός κανονισμός, πρέπει να υπάρχει πολιτική στήριξη. Δάλλως δεν γίνεται τίποτα. για την ε, διευκόλυνση της ε, κατανομής του κοινού οικονομικού κινδύνου. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση εδώ ότι τα σχετικά αποτελέσματα ήταν ε, πολύ καλά. Ίσως και λόγω της οικονομικής κρίσης να μην ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο αναμέναμε. Για την κυρία Χέρτσογκ έχουμε τα ποσοστά επιτυχίας. Είναι κειμενόμενα στους διάφορους τομείς με μεταξύ του 5% για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, κάτι που αυξήθηκε λίγο το μεταξύ, στο πρόγραμμα Άνθρωποι, People, βρήκαμε επίσης χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και χαμηλά και στο πρόγραμμα συνεργασίας, λόγω χάρη στις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές, αλλά και τις περιβαλλοντικές. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτά τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας είναι ότι αν σκεφτεί κανείς πόση δουλειά πρέπει να κάνει ένας ερευνητής για να ετοιμάσει μια πρόταση, μια υποψηφιότητα. Και μετά δει το ποσοστό επιτυχία που δεν ξεπερνά το 10%. Μετά θα κάνει την αίτηση. Αν λοιπόν τα δημοσιεύσουμε όλα αυτά, είναι σαν να ε, απογοητεύουμε του ανθρώπου που δεν κάνει υποβάλλουν την υποψηφιότητά του. Του αποθαρρύνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 12. Η εικόνα δεν είναι μαύρη ή άσπρη. Έχουμε έναν καθηγητή από την Εστονία, τον Τόιβο Άιματ στην Επιτροπή μα. και η Εστονία είναι σε τους υπόλοιπους 12 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι αρκετά επιτυχημένη. Όμω για τους υπολείπου υπάρχουν προβλήματα και το έχουμε συζητήσει διαμακρών. Τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα μα είναι ότι εφόσον το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο αφορά την αριστεία και την οικοδόμηση δυνατοτήτων, θα πρέπει να αναζητήσουμε αποτελεσματικότερη συνεργασία και με τα κοινωνικά ταμεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Για τις κοινέ πρωτοβουλίες είναι μια νέα μορφή συνεργασίας, όπου καταρτίζει και μια ατζέντα, μια σειρά προτεραιοτήτων η βιομηχανία ίδια. Δεν έχουμε αρκετή πείρα σχετικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω, γιατί η δραστηριότητες από τι οποίες ξεκινούμε δείχνουν ήδη τι θα ήθελε η βιομηχανία να συμβαίνει στο επίπεδο τη συνεργασίας. Απλώς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το είδους η συνεργασία. Και θίξατε και το θέμα της σχέσης κρατών μελών με τι ευρωπαϊκέ δραστηριότητες. Νομίζω απήντησα σε αυτό. Κύριε Γκίντης, όταν εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχα ασχοληθεί με την οδηγία για τη δικαιώματα ανταλλαγή εκπομπών. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα καταλήξουμε στην λογική να παίρνει κανείς τα κέρδη από, αυτήν, από αυτό το εμπόριο για να χρηματοδοτεί την έρευνα. Ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα σας, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ και να το σχολιάσω προς στιγμή. Πάντως ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι κάποιος θα επινοούσε κάτι τέτοιο. Για το EIT και CIP Αυτό δεν αποτέλεσε μέρος της αξιολόγησης. Όμως από τη στιγμή που παρουσιάσαμε την αξιολόγηση, ακούστηκαν ιδέες για ένα κοινό στατικικό πλαίσιο. Έναν τρόπο δηλαδή να συνδυαστούν όλες αυτές οι παράλληλες προσπάθειες. Νομίζω κάθε τέτοια προσπάθεια θα ήταν ε, ευπρόσδεκτη. Και θα ήταν και πολύ απλούστερο να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της καινοτομία και της έρευνας, εάν όλα τα συμπεριλαμβάναμε σε ένα κοινό πλαίσιο. Αλλά εδώ είναι δύσκολο να το υιοθετήσω αυτός προσωπική άποψη. Αυτό είναι περισσότερο δική σας άποψη και του Συμβουλίου. Και για τις ιδιωτικέ επενδύσεις επίσης, να πω ότι υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς δαπανάτε για αυτήν τη συνεργασία, αυτό το είδο συνεργασία από την ίδια τη βιομηχανία. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά για τα GTI, όμως ε, και για, την, για το εργαλείο κατανομής του κινδύνου τα πράγματα πάνε καλά. Ε, η συνεργασία αυτή σαφώ θα πρέπει να συνεχιστεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπατε. Οι στόχοι μας ε, δεν απέχουν πάρα πολύ. Μπορούμε να τους επιτύχουμε, απλώς παραμένουν κάποιες ελλείψεις και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα παγορευτικά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο. Όσο για τις υποτροφίες Μαρή Κιουρί, βεβαίως και είμαστε υπέρ όλου αυτού του συστήματος του Μαρή Κιουρί, όμως ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε και πόσο επιτυχημένο είναι το Κιουρί. Πόσοι από αυτές που πήραν χρήματα από το Μαρί Κιουρί πέτυχαν κάτι. Ή θα κάνουν αιτήσει για περαιτέρω χρηματοδότηση. Επίσης θέσατε το θέμα του συντονισμού των εθνικών ε, πολιτικών. Όπω είπα και νωρίτερα, συμφωνώ. Αυτό είναι ζήτημα, Μίζον ζήτημα. Επίσης, θέσατε το, το ζήτημα για το πώ θα πρέπει να έχουμε περισσότερους νέους ερευνητέ στο πρόγραμμα. Το Marie Curie, όπως λέγαμε, είναι σημαντικό για την πλαισίωση των νέων ερευνητών και για την αύξηση της κινητικότητας. Επίσης, θέσατε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνήσαμε γι' αυτό. Και έπειτα, το θέμα της ταχύτητας εκτέλεσης ε, από την πλευρά των διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής. Δεν το έχουμε καταμετρήσει, αλλά είδαμε ότι μπορούμε να βασιστούμε να βασιστούμε στην ε, συνεργασία των υπηρεσιών. Από τη στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν κάποιοι οργανισμοί, είδαμε να δυσκολεύονται στα αρχικά στάδια, αλλά κατόπιν να επιταχύνουν πάρα πολύ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Ο κύριο Τσουκαλά έθεσε το θέμα τη θέση τη ευρωπαϊκή έρευνα στο διεθνέ προσκήνιο πού βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή έρευνα σε σχέση με το τι συμβαίνει διεθνώ. Ο στόχο του 3% που είχαμε ορίσει στη στρατηγική τη Λισαβόνα και έχουμε κρατήσει για τη στρατηγική τη Ευρώπη το 2020 είναι στόχο που απέχουμε από το να το πετύχουμε. Κάτι σαν 5% νομίζω έχει ακουστεί κιόλα. Κάποιε χώρε στην Ευρώπη, όπω η Ιδία και η Φινλανδία, έχουν ξεπεράσει το 3%. Εάν όμω θέλουμε πραγματικά να είμαστε ανταγωνιστικοί, ιδίω σε σχέση με τι ΗΠΑ, οι άλλες ε, χώρες ε, την εφήλιο που χρηματοδοτούν την έρευνα και αυξάνουν και τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αυξήσουμε το στόχο του 3%. Να τον πετύχουμε και να πάμε και παραπέρα. Είναι άκρος αναγκαίο. Για το 4% που αναφέρατε, δεν είμαι βέβαιος ότι έτσι είναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Απλώς ε, υποστηρίζω ότι πρέπει να αλλάξει η ισορροπία μεταξύ πίστης, εμπιστοσύνης και κινδύνου. Διότι υποχρεωτικά θα χάσει κανείς χρήμα όταν είναι στην έρευνα, όχι γιατί γίνονται πάτες. Γιατί κάποιοι ε, άνθρωποι συχνά έχουν ιδέες, σκέφτονται πράγματα που δεν δίνουν κανένα αποτέλεσμα τελικά. Εάν ήξερε κανεί από πριν θα συμβεί, δεν θα πήγαινε στην έρευνα. Πρέπει να ρηψοκινδυνεύει κανεί κιόλα και να εμπιστεύεται του ερευνητέ όταν κάνουν μια πρόταση προγράμματο ότι πνευματικώ δεσμεύονται, είναι αφοσιωμένοι στο στόχο του. Αλλά είναι ερευνητέ, μην το ξεχνάμε. Πρέπει να τους αφήνουμε και ένα περιθώριο ελιγμού, αλλιώ δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει η έρευνα. Η κυρία Καρβάλιου τώρα. Είπατε αρχικά ότι όλα τα μέτρα απλούστευσης που ήδη διαθέτουμε θα πρέπει να εφαρμόζονται. Συμφωνούμε. 100%. Όσο για το θέμα του ERC δεν, έγινα, δεν έκανα πολλά σχόλια σχετικά όμως κάποιες από τις ιδέες για τη συνεργασία είναι πολύ σκόπιμες και για το μέλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Χρειάζεται κάποια σχετική πείρα για να μπορέσει κανείς να υποβάλει σωστά τις αιτήσει του για το πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε όμως ε, λόγω χάρη και ένα πρόγραμμα για να μάθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς καλύτερα να αξιοποιούν αυτά που προσφέρει το πρόγραμμα. Για την εμπορευματοποίηση, την ε, πλήρη αξιοποίηση, την ε, προσέγγιση της αγοράς, συμφωνώ απολύτως. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για την κυρία Γκουτιέρε Κορτίνε. Για το μορατόριο. Αυτό που είπα είναι ότι έχουμε επινοήσει πολλά, πάρα πολλά νέα εργαλεία για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα επινοητική και εφάνταστη. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε. Έχουμε το ERC, το E+, την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία και το καθεξής. Όταν μιλούσα για μορατόριο, για πάυση λειτουργία, δεν εννοούσε να σταματήσουν όλα αυτά να, να χρησιμοποιούνται. Πριν όμω επινοήσουμε κάτι καινούριο, α δούμε ήδη τι διαθέτουμε, τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Και μετά, με όλα αυτά τα εργαλεία, με όλα αυτά τα μέσα, με όλη αυτή τη δυνατότητα καινοτομία, δεν χρειάζονται άλλα νέα μέτρα. Θα δημιουργήσουμε σύγχυση μεταξύ των ερευνητών τη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μα δεν χρησιμοποιούνται όλα διαρκώς. Ε, χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα εργαλεία, να δούμε τι πάει καλά και τι όχι και να τα ξαναδούμε στο τέλος. Αλλά μην επινοείτε άλλα. Φτάνει. Προ στιγμή δεν χρειάζονται. Όσο για την καινοτομία και το τι γίνεται σε ποιο επίπεδο, η καινοτομία προφανώς είναι κάτι που λαμβάνει η χώρα σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι όλη η καινοτομία στις Βρυξέλλες, βεβαίω, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τι κάνουμε εδώ δημιουργεί τις συνθήκες πλαίσιο για την καινοτομία. Διευκολύνει την ε, ανάδυση της καινοτομίας στα κάτι μέλη. Ακόμη λοιπόν και αν η καινοτομία είναι κάτι που λαμβάνει χώρα σε εταιρείε των 100 μελών, προφανώς χωρίς δράση ευρωπαϊκή Εάν δεν είναι καλέ οι συνολικέ συνθήκε, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Συμφωνώ μαζί σα, η αριστεία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε όλα τα τμήματα του προγράμματο. Δεν σταθήκαμε ιδιαίτερα στο ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όμω προφανέστατα χρειάζεται εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Κάτι που ούτω ή άλλω διενεργείται σε όλη την Ευρώπη. Και μετά η κυρία Τόμσεν για την καινοτομία, τη μεταποίηση που αναφέρατε και τη σχετική βιομηχανία, Wirtschaft στα γερμανικά. Είναι ευρύτερο το θέμα. Για το τελευταίο σας σχόλιο είμαι ακριβώ της ίδιας άποψης. Η μεταφορά γνώσεων στι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ιδιαίτερη σημασία. Και κάποια τμήματα του προγράμματος αυτού, Όπω ανέφερα, τα Euro καταστήματα, τα Euro stores, μπορεί να είναι πολύ εξυπηρετικά στην συνδρομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ορίστε. Α, η κυρία Δελκαστήγιο. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Δεν μου φαίνεται δυνατό να συνδυάσουμε τις δύο συζητήσεις, γιατί τώρα συζητούμε για το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 7ου του πλαισίου και το επόμενο είναι η πρόταση που κάνει ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για την έρευνα. Δεν ξέρω, είναι λίγο συγκεχημένη η κατάσταση. Θα μπορούσαμε ίσως να περάσουμε αμέσως στη συζήτηση της πρότασης του κυρίου Οντή. Αλλιώς πότε θα το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται, δεν ταυτίζονται ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό το είπα προηγουμένω. Έκανα πρόταση γιατί είχαμε χρονικά προβλήματα, αλλά έχουν ζητήσει το λόγο 7. Αν μιλήσουν και οι 7, δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε το, το θέμα του κυρίου Οντί. Είτε θα διακόψουμε εδώ το σημείο 5 και θα περάσουμε μέσω στο 6 και θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε ε, με τη δεύτερη συζήτηση αυτά που είχατε να πείτε στην πρώτη. Αυτοί που θα μιλήσουν ακόμα, Τσικάου, Εκ, Έντσου, Βανίστε Ροϊ, Φόρτ, Βέμπερ και Ματίας. Μπορείτε να μιλήσετε. Περιμένετε, έχουμε μισή ώρα ακόμα και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Να μιλήσουν όλοι σύντομα, υπάρχει και αυτό. Αν μιλήσει ο καθένας ένα λεπτό, προλαβαίνουμε. Μπορεί και να προλάβουμε. Ένα λεπτό. Ελίνα Εκ. Παρακαλώ. Να το θέσουμε αυτό υπόψη της συνεδρίασης των συντονιστών που θα ακολουθήσει γιατί αυτοί που είναι τελευταίοι στον κατάλογο μπορεί να έχουν να πούν εξίσου σημαντικά πράγματα με τους πρώτους. Και δική σας δουλειά, Πρόεδρε, είναι να φροντίζετε να διανέμετε ε, ο χρόνος ίδια στους όλους. Εντάξει, να μην τσακωθούμε, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ πραγματικά φροντίζω να μιλάνε όλοι το ίδιο και να μιλάνε όλοι. Ορισμένοι δεν προλαβαίνουν να έρχονται ποτέ, ορισμένοι έρχονται μετά από ώρε. Άλλο θέλει να μιλήσει την ώρα που έρχεται. Αναβάλουμε το θέμα του τρει φορέ. Τι να κάνω τώρα. Ο καθένα ε, έχει μια νέα ιδέα για ακρόαση και όταν γίνεται η ακρόαση ο κόσμο δεν πατάει. Συγγνώμη που τα λέω έξω από τα δόντια. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο εδώ θα συζητούμε. Μόνο με τη σειρά. Έχουμε μια σειρά κατάλογο μιλητών, Αλλιώ πώ να προχωρήσουμε, τι άλλο να σα κάνω. Έχει κανένας μια πιο ευφυή πρόταση. Δύο προτάσεις ξέρω εγώ. Είτε τώρα θα μιλήσουμε πιο σύντομα, είτε δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε το θέμα του κυρίου αντί. Αν θέλετε και τα δύο. Προτάσεις. Μία πρόταση έκανα εγώ. Εγώ να μιλήσω και για τα δύο, αλλά θέλω να ακούσω απαντήσεις και για τα δύο μετά. Λοιπόν, πρόταση. Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια τη έκθεση ΟΝΤΗ και νομίζω ότι θα πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση για την έκθεση ΟΝΤΗ. Γιατί η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και συνδέεται με την έκθεση ΟΝΤΗ. Να συνεχίσουμε λοιπόν το σημείο 5 και να αναβάλουμε το 6. Αλλιώ πραγματικά δεν θα προλάβουμε. Καλώ. Τώρα θα κοιτάξουμε πώς θα προχωρήσουμε. Μπορεί, ε, προσπαθήστε να είστε σύντομοι όλοι ε, για να τα καταφέρουμε. Η κυρία Τσικάου πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Άνερμπερκ για την παρουσίασή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Είναι όντως σημαντικότατο. Επίσης θα πρέπει να ερευνήσουμε περισσότερο και να επενδύσουμε στην εφαρμοσμένη έρευνα, ιδιαίτερα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Παρατήρηση δεύτερη. Πριν από λίγα χρόνια συμμετείχα εγώ στην αξιολόγηση του 5ου τότε ακόμα προγράμματος πλαισίου και το συμπέρασμά μου στο οποίο κατέληξα είναι το εξής. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την προσπάθεια συγχρηματοδότησης που πρέπει να καταβάλει μια μικρομεσαία επιχείρηση με την προσπάθεια έρευνα στην οικονομική μιας μεγάλης εταιρείας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μια μικρή μεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να ε, εξασφαλίσει την ίδια συγχρηματοδότηση. Και δεν θα πρέπει αυτό να είναι εις βάρος των επιχειρήσεων, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν όπως οι μεγάλες εταιρείες. Και τέλος, όταν κανείς κάνει μια ταξινόμηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν άλλη μεταχείριση μικρές εταιρείες. Οι μεγάλες δεν έχουν πρόβλημα χρηματοδότησης ενός προγράμματος. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που να προσανατολίζεται αποκλειστικά στις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης, να είναι και αυτές διαφοροποιημένες, διότι Ανάλογα με την εκάστοτε πηγή χρηματοδότησης, όταν υποβάλλεις μια αίτηση, τα κριτήρια που καλείσαι να καλύψεις είναι πολύ διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό. Αν θέλει κανείς να έχει όσο γίνεται περισσότερη χρηματοδότηση, θα πρέπει να πληρεί διάφορα κριτήρια, πάρα πολλά. Και δεν μπορεί να υποφελείται από τις νέες πηγές χρηματοδότησης. Αυτά προτείνω, λοιπόν. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε μια σύγκληση μεταξύ αυτών των κριτηρίων αξιολόγησης και χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Λίνα Εκ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, συγχαρώ την ομάδα των εμπειρογνωμών για την ποιότητα της έκθεσης και της εργασίας γιατί αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα που ε, κατατέθηκαν τον τελευταίο καιρό στην Επιτροπή μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ε, θα είναι καθοριστικό όχι μόνο για την διάμεση αναθεώρηση αλλά και για τον προγραμματισμό και τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα υπαριθμών 8. Όσον αφορά τώρα το συντονισμό ανάμεσα στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και άλλα εργαλεία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, φέρει μεγάλη ευθύνη και θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις για το πώς ε, ακριβώς μπορεί να γίνει ο συντονισμός σε τομείς όπως η εφαρμογή, η χρηματοδότηση, IPR και άλλα πρακτικής φύσεως ε, θέματα τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή τα γραφειοκρατικά εργαλεία δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και κατά την άποψή μου όπως σας είπα γι' αυτό φταίνει λένε οι Γενικέ Διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την επιτυχία και την αποτυχία, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Έρευνα πρέπει να ανακοινώνει και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες γιατί πρέπει να μπορούμε να ε, ισχυριστούμε, να επιχειρηματολογήσουμε γιατί χρειαζόμαστε κονδύλια για την καινοτομία ε, να δείξουμε το τι, ε, τα τι προκάλεσαν τα προγράμματα τα θετικά του αποτελέσματα και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει κανείς μόνος. Θα πρέπει να περάσει ολόκληρες μέρες στο διαδίκτυο και σε συναντήσεις με τους αρμόδιους. Κατόπιν, όσον αφορά τα νέα εργαλεία. Ένα από τα προβλήματα με την πρωτοβουλία, ε, την κοινή πρωτοβουλία είναι ότι αυτό το εργαλείο στην αρχή εκπονήθηκε ως κάτι το καινούριο, αλλά ε, τελικά απορρίφθηκε ως, ε, και υποβαθμίστηκε ως ε, διοικητικός ε, κανονισμός. Ίσως λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει το δικαιοστάσιο. Τα νέα εργαλεία, με τα νέα εργαλεία, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν βρίσκουν κάτι που να λειτουργεί και γι' αυτό προχωράνε παραπέρα. Δεν ξέρω αν το δικαιοστάσιο, το moratorium είναι ίσως τη λέξη που να εκφράζει τις επιφυλάξεις ομάδας. Και τέλος, όσον αφορά στη συμμετοχή και πιο συγκεκριμένα για τη βιομηχανία βλέπουμε ότι το επίπεδο συμμετοχής ε, της βιομηχανίας περιορίζεται ε, συνεχώς στα διάφορα ερευνητικά ε, προγράμματα. Και αν συγκρίνουμε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κανδύλια που δίδονται για την έρευνα είναι περίπου τα ίδια. Αν προσθέσει, από το δημόσιο τομέα, αν προσθέσει όμως και τα κονδύλια του ιδιωτικού τομέα, βλέπουν ότι η διαφορά είναι τεράστια. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για το πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν συζητούν περισσότερο τα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πραγματικά τα χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, ε, πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση που έχουμε λάβει και είναι δυσάρεστο το ότι ε, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές οι αρχές και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα μιλήσουμε για τον έλεγχο. Σχετικά με το άρθρο 185 εγώ διαπραγματεύτηκα το πρόγραμμα Bonus που αφορά την έρευνα για τη Βαλτική. Και Όσον αφορά την κοινή ε, πρωτοβουλία τεχνολογίας, εγώ διαπραγματεύτηκα για τους καθαρούς ουρανούς, ε, το Clean Sky και αυτό ισχύει και για το άρθρο 185. «Επαρχόμαστε συνεχώς την απλούστευση και την αποτελεσματικότητα. Και τέλος κύριε Πρόεδρε ε, θα μου επιτρέψετε κάποια σχόλια για το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Υπήρξε μία δήλωση από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο το ίμιση των εσόδων από τις ε, ανταλλαγές αυτές να δαπανάτε σε έρευνα για την πράσινη τεχνολογία και συναφείς τομής. Ελπίζω λοιπόν και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και το 50% των εσόδων από αυτές τις ανταλλαγές να το χρησιμοποιήσει όπως έχει υποσχεθεί. Μπορείτε να δείτε τις δύο ανακοινώσει της Κομισιόν την Τρίτη. Η μία αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και η άλλη ε, το χάρτη πορείας μέχρι το 2050 και θα καταλάβετε αν τα δείτε όλα αυτά γιατί πρέπει να γίνουν αυτά που μόλις σας προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριο Σέντσου. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το προσκεκλημένο μας για την έκθεση και την παρουσίαση της αξιολόγησης εδώ. Η μεγάλη πλειονότητα των όσο ήθελα να πω καλύφθηκε από τους συναδέλφους. Οπότε εγώ θα αναφέρω ένα και μόνο θέμα που πραγματικά με προβληματίζει και με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ευρώπης των 15 και της Ευρώπης των 12 στη συνέχεια. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχής τους στα ερευνητικά προγράμματα των νέων χωρών μελών. Μπορεί να απαντήσει παρακαλώ ο, ο κύριος Άνενρπερκ. Πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά, πώς μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή τους. Βεβαίω, οι κυβερνήσει των κρατών αυτών δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ, ούτε προσπαθούν να καταλάβουν τη σημασία που μπορεί να έχει έρευνα και καινοτομία. Χάρη στην έρευνα και την καινοτομία θα μπορούσε να μειωθεί μέχρι και το ποσοστό της φτώχειας. Πώς μπορούν να στηριχθούν λοιπόν οι νέες χώρες για να συμμετέχουν περισσότερο στην έρευνα κατά την άποψή μου, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και για την υποδομή. Κατά τη μεταπολίτευση, τη μετάβαση από το κομμουνισμό ε, στη νέα κατάσταση, ε, καταστράφηκε πολύ ε, μεγάλο τμήμα της παλιάς ερευνητικής υποδομής που είχαμε και είναι τελείως απαρχιωμένη. Πλην όμως το δυναμικό υπάρχει το οποίο δυναμικό αυτό δεν το εκμεταλλεύονται, δεν το αξιοποιούν τα παλιά κράτη-μέλη. Από τη Ρουμανία, ας πούμε, η συντριπτική πλειονότητα των νέων ερευνητών πηγαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτυχθούν. Ο κύριος Φανίσερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ εκτιμώ ε, την έκθεση αυτή. Ε, ε, κοιτάω τη σύνοψή τους και τη ε, από τη σύνθεσή τους. Είναι Φιλανδοί, Εστονός, Βέλγος. Πώς ε, έγινε αυτή η σύνθεση της Επιτροπής αυτής. Είναι ε, όλες αυτές οι χώρες που βρέχονται από τη θάλασσα. Γιατί τους βοηθάει ο θαλάσσιος αέρας, η άβρα. Πώς τους επιλέγετε. Είναι τελείως σύμπτωση ότι όλοι προέρχονται από χώρες της Βαλτικής, της Βορείου Θάλασσας ή του Ατλαντικού. Εσείς ήταν πρόεδρος. Δεν θα μπορούσατε να είχατε πει ότι ε, όχι έτσι. Δεν ξέρω γιατί, πώς ε, ε, αυτή η γεωγραφική αλληλεγγύη στην Ένωση. Είναι τυχαίο που έχει έτσι η σύνθεση και είναι ε, κάποια ανισορροπία. Και η κυρία Έκτο ρώτησε ε, είναι ένα θέμα αγαπημένο αυτό ότι επενδύουμε ε, στην, ε, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλο λόγο εκεί. Στα διαρθρωτικά ταμεία, βεβαίως, στα νέα κράτη-μέλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο τα περιφερειακά ταμεία για να ε, βελτιώσουμε τις υποδομές. Ε, έρευνα, όπως είπατε τώρα, 40 ε, δισεκατομμύρια στην παρούσα προγραμματική περίοδο αναφέρονται, αφιερώνονται εκεί από τα διαρθρωτικά ταμεία για την έρευνα. Το έχετε ψάξει αυτό? Έχετε μερικά στοιχεία αριθμητικά? Πού πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια, γιατί είναι και περίπου μόνο καλλιέργεια, γιατί μοναδική ε, αναφοράς. Αυτό το Facility Fund ε, είναι μια δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων. Αυτό που θα με ενδιαφέρε είναι να έχουμε υποδομές. Αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις που θα πρέπει να τονώσουμε γιατί δεν επενδύουν οι άλλοι σε αυτές. Αυτό πόσο σχολιάζετε σας. Η κυρία Φόρτ. Um, thank you. Um, thank you for starting by speaking about excellence and so positive. Ε, κοιτάξτε, θα ήθελα να πω καταρχήν ε, ε για την αριστεία. Εγώ είμαι σαφώ υπέρ, έχω, είδα ότι χρονοτοδίκαμε πολλά ε, προγράμματα που έχουν σχέση με την αριστεία. Ε, η Ευρώπη πρέπει να ζητήσει τον χώρο της ε, στην έρευνα μέσα στο ευρύτερο σκηνικό, γιατί εκεί κινδυνεύουμε να είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί. Και σε ευχαριστώ πολύ που προσπαθείτε να μας ε, στρέψετε προς τις μεγάλες ε, προκλήσεις, γιατί πραγματικά εκεί πρέπει να δαπανώνται τα περισσότερα κονδύλια. Για μένα η απλούστευση είναι καθοριστική σημασία και δεν μπορώ ε, και όσοι εργαστήκαμε την έκθεση Καβάλιο, πραγματικά ε, είδαμε ότι υπήρξαν πάρα πολλέ συστάσει για την απλούστευση και δεν έγινε τίποτα τελικά. Και ο λόγο ε, που αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό είναι ότι αν δεν εφαρμόσουμε την απλούστευση θα υπάρχουν συνεχώς και άλλα προσκόμματα. Γιατί δεν συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, γιατί τα πράγματα είναι όλο και πιο περίπλοκα και ξέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι η γειτονική ας πούμε κατεστράφη, πτώχευσε γιατί δεν πήρε τα κονδύλια που της είχαν υποσχεθεί. Η απλούστευση λοιπόν είναι καθοριστική σημασία. Η δική μου χώρα είναι εκτός ευρωζώνης ε, και ξέρετε υπάρχουν πολλά θέματα σημαντικά ε, που αφορούν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ε, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τόσο περίπλοκα. Αν δεν έχουμε όλες τις διαβουλεύσεις για τα συναλλαγματικά, τα πράγματα ήταν πιο απλά. Για μένα λοιπόν η απλούστευση είναι καθοριστική σημασίας και διερωτώμε για το κατά πόσο μπορεί να αναζητηθεί ε, κάποιος συμβιβασμός ε, για μικρά προγράμματα. Πράγματι ε, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους που να είμαστε διατημένοι να αντιμετωπίσουμε. Όμως όσο αυξάνονται τα κονδύλια θα πρέπει να εμπλέκεται λιγάκι και η Κομισιόν. Να υπάρχει ένας συμβιβασμός ανάμεσα στους μικρούς τις μικρές επιχειρήσεις και ε, στα, στις μεγάλες. Εγώ ε, θεωρώ ότι η χρηματοδότηση, ε, το εργαλείο χρηματοδότηση κινδύνου εστιάζεται σε ορισμένες χώρες, είναι πολύ στοχευμένο σε ορισμένες χώρες και διαρωτώ με κατά πόσον εις αυτό οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρείται περισσότερο η τράπεζα της Ευρωζώνης ή μήπως απλά το εργαλείο αυτό δεν έχει διαφημιστεί αρκετά στα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι ας πούμε στη δική μου τη χώρα το εργαλείο αυτό ε, είναι σχεδόν ανύπραπτο, κανείς δεν το ξέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος επιστήμονες που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν να ζητήσουν χρηματοδότηση. Πράγματι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουμε ε, χώρες ε, που δεν έχουν προχωρήσει ερευνητικά παιδεία και θέματα να προχωρήσουν, να μην υπάρχει στενοπός. Τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με καλύτερο τρόπο. Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα ταμείο, δεν είναι διαρθρωτικό, ένα ταμείο που προάγει την έρευνα και την καινοτομία. Δεν πρέπει αυτή την ε, αριστεία ε, να την θέτουμε σε κίνδυνο. Θέλουμε να υπάρχουν διευθυντικά ταμεία, αλλά θέλουμε και να ε, διοχετεύονται με τον καλύτερο τρόπο. Έχω και κάποια άλλα σχόλια να κάνω. Είναι καλή έκθεση γενικές γραμμές και θα πρέπει εν κατακλείδη να είμαστε και ικανοποιημένοι με την έκθεση που κατατέθηκε. Ο συνάδελφος κ. Βίμπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κ. Βεμπέρ, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα μόνο σημείο από αυτά ε, που είπατε. Υπάρχει η δυνατότητα να διορθώσουμε το τα βασικά μειονεκτήματα που έχουμε στην ευρωπαϊκή έρευνα ε, τρεις φορές απλούστευση και στο διοικητικό και στο γραφειοκρατικό άχθος, διατηρώντας τις ίδιες δομές. Διάβασα την έκθεση ε, με ενδιαφέρον του φίλου μου καθηγητού Ιβμενή, που ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και προτείνει μία ε, αναθεώρηση, μεταρρύθμιση ε, των δομών, των υποδομών. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό. Είναι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που είναι εκτελεστικό όργανο, εκτελεστικός οργανισμός και προτείνει να γίνει ανεξάρτητο ε, νομικό πρόσωπο με δυνατότητα λήψης αποφάσεων και που να είναι άμεσα αρμόδιο και για την επιστημονική στρατηγική αλλά και για τη διοικητική διαχείριση. Θα ήθελα την άποψή σας για την έκθεση αυτή η μενή και γενικά την άποψή σας επίσης για αυτή την πρόταση να αλλάξουμε τις δομές, διότι... Πώς να το πω... Εάν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ρυθμίσεις και μάλιστα τις πολλαπλασιάζουμε, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα βασικά αυτά μειονεκτήματα που έχουμε εντοπίσει εδώ και καιρό, αλλά ε, λίγο μόνο έχουμε προχωρήσει στην επίλυσή τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα όσα μας υπέβαλε. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά για τη μελέτη μας και όλη αυτή η προσπάθεια για την αναθεώρηση των ε, διαφόρων στοιχείων του προγράμματος πλαισίου. Όχι μόνο γιατί μιλάμε και για ένα πρόγραμμα με υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης, με δημόσια κονδύλια και απόψη διεθνή μάλιστα, αλλά που θα έχει και πολύ σημαντικές επιπτώσεις για όλους. Ήθελα λοιπόν ε, να κάνω κάποια πρώτα σχόλια και να θέσω και κάποιες ερωτήσεις. Ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με την απλούστευση και τα όσα γνωρίζουμε για τον ε, πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση των ερευνητικών εργαλείων. Να πω ότι ως πρώην ερευνήτρια που εργάστηκα στο 5ο και έκτο ο πρόγραμμα πλαίσιο με διάφορα επιμέρους προγράμματα, πολλές φορές αισθανόμασταν σαν πειραματόζωα, σαν ποντίκια σε ένα πείραμα που κάθε φορά μας επέβαλαν ε, και μας επέβαλαν τη χρήση νέων εργαλείων και νέων μέσων. Ήμασταν εμεί οι ίδιοι το αντικείμενο του πειράματο. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που υπήρξαν θετικά αποτελέσματα εντωμεταξύ και η έκθεση Καρβάλιο είναι πολύ σημαντική σχετικά και πολύ εύστοχη. Είναι μια έκθεση που θα τη συζητήσουμε ούτω ή σε μια άλλη φάση, μετά από την έκθεση του κ. Ντί. Εδώ τρει παρατηρήσει λοιπόν σε σχέση με όλα τα κοινά ζητήματα που μα απασχολούν. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για την έρευνα. Άρα η χρηματοδότηση είναι ευρωπαϊκή. Πολλές φορές νομίζω ότι παραμελούμε τις διαφορές που υπάρχουν εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Η δομή αυτή για το πρόγραμμα πλαίσιο διαθέτει κάποια μέσα συνεργασία, συγκεκριμένα άτομα, δυνατότητες, όλα αυτά είναι γνωστά θεωρητικά. Όμως, η αποτίμηση πρέπει να γίνεται εις βάθος, να μπαίνουμε δηλαδή στις λεπτομέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ερευνητικό χώρο τη Ευρώπη θα πρέπει να είναι ισχυρό, αλλά προηγουμένω για να περάσουμε στο διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να δούμε τι εσωτερικέ μα διαφορέ. Τα μέσα οργάνωση και έρευνα και τα διάφορα εργαλεία δεν φτάνουν στο 100% των δεκατοτήτων του ακριβώ επειδή υπάρχουν αυτέ οι εσωτερικέ διαφορέ. Και οι δυσκολίε τη χρηματοδότηση, όπω είπε και ο συνάδελφο προηγουμένω, κάποιε φορέ ε, φτάνουμε στο 50% για του πιο ενεργό συμμετέχοντες από όλη τη συμμετοχή. Και δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες, ούτε τα ακαδημαϊκά κέντρα, ούτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ούτε τα ερευνητικά, ούτε αναγκαστικά όλοι οι φορείς της βιομηχανίας. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να δούμε το τους 50 καλύτερους και της Ευρώπης και της Γερμανίας, της Γαλλίας, αλλά λόγω χάρη πόσοι από αυτούς είναι από την Πορτογαλία σε αυτό το 50. Εδώ το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Όπως και το ότι θέλουμε να ενισχυθεί η συνοχή στην Ευρώπη. Ένα εργαλείο είναι, αυτό το εργαλείο μάλλον της είναι πολύ σημαντικό και για τη συνοχή. Δεύτερη παρατήρηση. Με τα πρόσωπα τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τους ανθρώπους, γιατί δεν θέλω να σταθώ στα μέσα και τα εργαλεία. Στα πρόσωπα λοιπόν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, έχει αυξηθεί κινητικότητα, έχει αυξηθεί η διάδοση των μέσων χρηματοδότηση, όπως η ο Μαρή Κιουρί. Όμως εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το εργαλείο είναι πολύτιμο όχι μόνο για τη σταδιοδρομία των ερευνητών, αλλά και ως ε, μέσω ε, σταθεροποίησης ε, σταδιοδρομίας θα ήταν σημαντικό να αντιμετωπίζεται. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έρευνα στην Ευρώπη πολλέ φορέ βασίζεται σε επιστημονικό έργο προσωρινό, που διέπεται από την προσωρινότητα. Είναι πολύ άνισε οι συνθήκε εργασία στην Ευρώπη και σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου που έχουν ανάλογα ερευνητικά προγράμματα. Και μια τρίτη παρατήρηση με την οποία θέλω να κλείσω είναι οι προτεραιότητες. Γνωρίζω ότι ο ορισμός των προτεραιοτήτων είναι ορισμός πολιτικός, πολιτικού χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να παραμελούμε μια απαραίτητη αποτίμηση που χρειάζεται είτε ενδιαμέσως είτε μετά τη λήξη του κάθε προγράμματος πλαισίου και πριν το επόμενο. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι, ποιοι είναι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά και αν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Διότι α πούμε ότι ένα μεγάλο μέρο τη χρηματοδότηση πήγε στη βιοτεχνολογία γιατί εκεί θέλαμε να πάει, μετά στην ανοτεχνολογία, μετά στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Υπήρχε ε, αύξηση για την άμυνα. Αρωτώ όμω, τελικώ τα αποτελέσματα ποια είναι. Γιατί γνωρίζω ότι αυτέ είναι πολιτικέ προτεραιότητε. Μεν, αλλά θέλουμε τουλάχιστον κάποια δεδομένα, κάτι να μας δοθεί, ώστε να καταλάβουμε εάν ως προς την αξιολόγηση οι αρχικοί προσανατολισμοί, οι πολιτικοί προσανατολισμοί για τις προτεραιότητες έδωσαν τελικά πρακτικά αποτελέσματα ή απλώς αλλάζουμε περιοχή και τομέα ανάλογα με τη μόδα. Και εδώ να θυμίσω και την έκθεση του συναδέλφου Οντί, με αυτό το συσχετισμό θέλω να κλείσω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο που μα υπέβαλε, το σημείο 30, εκεί που λέει ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να καλύψουμε την αξιολόγηση που μας λείπει τα τελευταία χρόνια και για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χρηματοδότηση που τόσο πολύ μας λείπει. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω ξανά τον κύριο Άνερμπεργκ να κάνει μια προσπάθεια να απαντήσει σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μπορεί να μην μιλήσω πάνω από τέσσερα λεπτά. Ε, κυρία Τεκάου, ε, όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατά 75% και μεγάλες επιχειρήσεις κατά 50%. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά προγράμματα μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ είμαι λιγάκι επιφυλακτικός, διότι πιστεύω ότι εδώ το σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κύριε Ικ, Ικε, ε, κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή και κάποιες προς εμένα που αφορούν ε, στις δυσκολίες για τη χρηματοδότηση. Αν λοιπόν ε, υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για όλους, νομίζω ότι τότε ε, θα είχαμε επιτύχει κάτι το ιδιαίτερα επικοδομητικό. Και όπως αναφέρατε, δεν, μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώ πόσα κονδύλια δόθηκαν για το GTI, αλλά αυτό ε, που είπατε εσύ είναι αλήθεια. Ε, Φίξατε την, ε, το χάσμα επίση ανάμεσα στους 12 και τους 15. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα τα κρατη κράτη-μέλη πρέπει μόνα τους να θέσουν τις ερευνητικές τους προτεραιότητες και μετά μπορεί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διευθυντικά ταμεία για να αυξήσουν τους πόρου. Όσον αφορά τώρα τη σύνθεση ομάδας, όπως ε, θα ακούσατε, ε, η σύνθεση ομάδας είναι κάπως βόρεια, υπάρχει όμως ε, ένα όνομα που είναι παραπληκτικό, η Σουζάνα Μπόρες, που δουλεύει στην Κοπενχάγη, αλλά αυτή είναι Ισπανίδα. Πάντως πράγματι δεν υπάρχει ισορροπία. Να σε εξηγήσω όμως ακριβώς τι έγινε. Πρώτον, όταν εμένα μου ζήτησαν να αναλάβω αυτό το ρόλο, του είπα ότι εμένα δεν με νοιάζει ποιο ε, θα βρίσκεται στην ομάδα. Εξ όσων γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει τις δικές της απόψεις όσον αφορά το βορρά, τους άνδρες, γυναίκες, κάποιες συγκεκριμένε ε, εγώ είπα ότι θέλω να έχουμε 7 συναντήσεις και όσοι ε, θα συμμετάσχουν να παρίστανται τουλάχιστον 5 φορές. Και με αυτό το αίτημα χάσαμε αρκετούς. Ε, το πώς τελικά τα βολέψαμε. Ε, πρώτον, από την Αυστρία, τη Γαλλία και από άλλου ε, μα έστειλαν αναπληρωτέ. Εμεί είμαστε αναχτές, ανοιχτοί σε οποιονδήποτε από την Ευρώπη που θέλει να εκφράσει κάποια άποψη. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι ακόμα και αν αυτό δεν σα μοιάζει ιδιαίτερα ισόρροπο, η σύνθεση δηλαδή, εμεί ε, δουλέψαμε με διαφάνεια, ακούσαμε τι απόψει όλων, ε, ό,τι μα είπαν από του οργανισμού, από τι διάφορε χώρε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη και η σύνθεση είναι ισορροπημένη. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δομές και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κινδύνου, ε, αυτό που βλέπουμε στην, ε, σε μία από τις συστάσεις μας είναι ότι Κατά την άποψή μας, ε, το εργαλείο αυτό, χρηματοδότηση κινδύνου, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο ως προς τη χρηματοδότηση της υποδομής στην Ευρώπη. Και δεν έχει τύχει μέχρι τώρα σωστή εκμετάλλευση. Κυρία Φόρτ, συμφωνώ απόλυτα βέβαια με αυτά που είπατε για την απλούστευση που είναι και παραμένει το κλειδί της όλης ιστορίας. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που είπατε για το T.A.E αλλά είναι κάτι ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Τώρα, όσον αφορά το SSF, δεν ξέρω αν σε ορισμένες ε, χώρες ε, ε, είναι πολύ στοχευμένο. Οι άνθρωποι μας έρευνα μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτό το εργαλείο. Ο κύριος Βίμπα, πράγματι και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να απλουστεύσουμε τις δομές. Ίσως θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, πρόταση με την αξιολόγηση του ERC και να γίνει αυτό ε, περισσότερο ανεξάρτητο. Δεν το θίξαμε αυτό, απλά καταλήξαμε ε, στο ότι αυτά που κάνει το ERC είναι πράγματι εργασία ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου. Προς εσάς κυρία Ματίας, βεβαίως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και αν δείτε τις, ε, ε, τους, και, την ε, Αμερική νομίζω θα, θα ήθελα να πει ο μιλητής. Πάντως πρέπει να δούμε γιατί ξεκίνησε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Βεβαίως αριστεία στην έρευνα, αλλά και μέσα από την αριστεία στην Ευρώπη μπορεί κανείς να προάγει και την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό. Και νομίζω ότι ε, τέλειωσε ο χρόνος μου, δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Κύριε Άνερβαχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο που ήρθατε, δεύτερον που μας ενημερώσατε με τέτοια λεπτομέρεια και χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει αρχικά μια μισή ώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ανάγκη για διευκρινήσεις και μας δώσατε και πάρα πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκληρώνεται εδώ αυτό το σημείο της μέσης διάταξης. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Και μόλις άκουσα ότι η κυρία Φόρτ την τρίτη απουσιάζει για το θέμα της. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να μεταθέσουμε την έκθεση του κυρίου Οντή για αύριο, αν συμφωνείτε. Και την Τετάρτη της κυρίας Φόρτ. Εάν συμφωνείτε, εντάξει, αν, περάσει εύκολα, αν χρειάζεται συζήτηση, δεν θα την κάνουμε τώρα. Ε, εγώ θεωρώ ότι αύριο εκεί που θα έπρεπε να είχαμε συζητήσει την ε, έκθεση κυρίας Φόρτ, θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Οντή, εμβόλυμα, και την Τετάρτη το θέμα της κυρίας Φόρτ. Διαφωνείτε, επιφυλάξει έχετε. Τι ώρα, δεν ξέρω τι ώρα, θα εξαρτηθεί από το πώς θα μιλήσουν, θα μιλήσουν πριν από την έκθεση αυτή. Δεν ξέρω, πρέπει να το κοιτάξουμε. Ποια είναι η καλύτερη ώρα για την έκθεση Φόρτ, την Δετάρτη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά... Δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ πριν τις 12 το μεσημέρι, γιατί συμμετέχω συνεδριάσει των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα πρέπει να σεβόμαστε και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εκεί θα πάω δηλαδή, εδώ θα είμαι. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο χώρο και να μου πείτε εσείς πότε να έρθω, πώς θα προχωρήσει η μερίσια διάταξη, αν προλαβαίνω. Θα ήταν καλό για τους και αν είναι όλοι εδώ και την Τετάρτη. Αλλιώς μετά τις 12 είμαι εδώ. Θεωρώ ότι η γραμματεία θα σας ενημερώσει όλους πότε θα γίνει αυτό την Τετάρτη. Άλλαξε τώρα η μερίσια διάταξη. Εκ των υστέρων ε, θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι και οι απόντες. Λοιπόν, πρώτον, αύριο στη θέση ε, του 12 θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Οντή και μετά να δούμε πότε την Τετάρτη ε, ε, θα μπει η έκθεση κυρίας Φόρτ. Τι ώρα. Συμφωνείτε. Εντάξει, τις λεπτομέρειες θα τις λύσουμε. Ευχαριστώ. Λήξη συνεδρίαση παρακαλώ να παραμείνουν οι συντονιστές. <laughs>